Dear colleagues, uh, to start. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχει έρθει η ώρα να ξαναρχίσουμε. Ε, καλωσορίζουμε τον Επίτροπο ε, κύριο Βέλα. Θα ήθελα αμέσω να αρχίσουμε τη συζήτηση μαζί του, διότι μεταξύ άλλων έχουμε χρονική πίεση. Ο Επίτροπος πρέπει να φύγει στις 5 και ζητήσαμε από τον Επίτροπο να έρθει στις 4 εδώ, μεταξύ άλλων διότι πρέπει να συζητήσουμε μαζί του θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική βιοπικιλότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ως συνήθως θα αρχίσουμε με μια εισαγωγική τοποθέτηση ε, από πλευράς Επιτρόπου. Θα ακολουθήσει ένας πρώτος γύρος ερωτήσεων από τους ε, συντονιστές και ο Επίτροπος θα απαντήσει ε, συλλογικά και μετά θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος για τα μέλη της Επιτροπής. Παρακαλώ, θα δώσω το λόγο στον κύριο Βέλα για την αρχική του τοποθέτηση και θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ Τζοβάνι. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, καταρχάς σας ευχαριστώ που με υποδέχεστε και πάλι στην Επιτροπή σας για να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα από ε, της έκθεσης ε, για την κατάσταση της φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πριν από λίγες εβδομάδες παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιστροπή. Είναι βασικό ε, αυτό έγγραφο στο check-up που κάνουμε για τη ε, νομοθεσία για τη φύση και την ενδιάμεση αναθεώρηση για τη στατηγική βιοπικιλότητα. Επιτρέψτε μου σύντομα να σας ενημερώσω και για τα δύο θέματα. Είχα πολύ καλές ε, συζητήσεις το Μάιο με τους Υπουργούς στο Άτυπο Συμβούλιο Περιβάλλοντος και είναι μια καταπληκτική ευκαιρία αυτή που έχω σήμερα να ακούσω και τις δικές σας απόψεις για αυτά τα θέματα. Ας αρχίσουμε λοιπόν από την έκθεση για την κατάσταση της φύσης. Θα πρέπει να είμαστε πολύ ε, περήφανοι. Ε, είναι μια μελέτη για τους οικοτόπους και τα είδη μετά από γόνιμη και στενή συνεργασία μεταξύ ε, κρατών μελών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ιδιαίτερα θα ήθελα να τονίσω και να εξάρω το σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ε, που συνέλεξε και ανέλησε τα στοιχεία. Τι μας λέγουν λοιπόν αυτά τα στοιχεία και ποιες είναι οι συνέπειες και τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξαγάγουμε. Οι Ευρωπαίοι έχουν διαμορφώσει το πεδίο και επηρεάσει ε, τη μοίρα της φύσης, το τοπίο μάλλον, και έχουν επηρεάσει τη μοίρα της φύσης για αιώνες. Το τελευταίο αιώνα όμως ε, έχει ενταθεί η γεωργία, έχουν αναπτυχθεί υποδομές, έχουν διευρυνθεί και επεκταθεί οι πόλεις, ε, αλλά και οι ρήπανση έχει αυξηθεί και ο φόρος που εκλήθη να πληρώσει η φύση ήταν πάρα πολύ βαρύς. Η αφετηρία για την νομοθεσία μας λοιπόν σχετικά με τη φύση ήταν να σταματήσουμε οποιαδήποτε περαιτέρω απώλεια και παρακμή και να ε, επανέλθουν ε, όσο γίνεται στην αρχική τους μορφή, οι κότοπη και η φύση, γιατί στο κάτω-κάτω εξαρτώμεθα απολύτως από αυτά. Είναι ε, το έργο αυτό πάρα πολύ απαιτητικό και ε, ε, όλα αυτά παραμένουν σήμερα πάρα πολύ επίκαιρα, θα συμφωνήσετε μαζί μου. Η φύση ωστόσο δεν ανταποκρίνεται πάντα με ταχύ ρυθμού στα μέτρα που εμείς λαμβάνουμε. Τα ε, καλά νέα είναι ότι η εφαρμογή των οδηγιών μας για τη φύση έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Για παράδειγμα, ε, ήδη όπως είναι οι ενιδρίδες ξαπλώνονται και πάλι παντού στην Ευρώπη. Ορισμένα Φτηνά επίσης επανέρχονται και τα έργα από το πρόγραμμα LIFE για την αποκατάσταση δύο τόπων και οικοτόπων ε, αρχίζουν να αποδίδουν πλήρως. Το δίκτυο Natura 2000 προστατευμένων περιοχών που είναι η ραχοκοκαλιά της νομοθεσίας μας ήταν ε, ε, κάτι στο οποίο εστιάσαμε και για την έκθεση αυτή πόσο αποτελεσματική είναι. Ε, και άλλα καλά νέα σας έχω. Είδαμε και διαπιστώσαμε ότι το δίκτυο έχει ε, μια σημαντική επίπτωση σταθεροποίησης ε, σε οικοτόπους και σε είδη που ακόμα είναι σε δυσμενή κατάσταση. Επίσης, κάποια είδη πτηνών που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές εμφανίζουν τάσεις πιο εθαρρυντικές από άλλα είδη. Ωστόσο φυσικά τα πράγματα απόρο απέχουν από την ιδεώδη κατάσταση. Χάνουμε ακόμα βιοπικιλότητα και ένα σημαντικός αριθμός ειδών και οικοτόπων ε, εξακολουθούν να είναι σε ε, ύφεση. Είναι γεγονός ότι οι επενδύσεις στη φύση όπου έγιναν έχουν αρχίσει να αποδίδουν καλά και ε, σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση πληθυσμών ειδών και οικοτόπων αλλά και το οικοσύστημα και τις υπηρεσίες που παρέχει ένα οικοσύστημα στην κοινωνία γενικότερα. Ωστόσο, δεν είναι αρκετή η πρόοδος για να πούμε ότι φτάσαμε στους στόχους που είχαμε θέσει ε, στη στρατηγική μας για τη βιοπικιλότητα. Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα τώρα για τη φύση. Ε, η συνολική εικόνα είναι σαφής. Για την ε, χερσαία πτυχή ε, το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η γεωργία. Για τη θάλασσα ε, η χρήση των θαλασσίων πόρων και η ρήπανση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ε, βεβαίως αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι κάτι που μας πλήσει πραγματικά, αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε ποιες είναι οι καλύτερες λύσεις για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα τα οποία πολύ καλά γνωρίζουμε. Ένας βασικός ε, παράγων είναι η χρήση των κοινοτικών κονδυλίων. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες για να υποστηριχθεί η διαχείριση και η αποκατάσταση του δικτύου Natura 2000. Ε, δεν έχουν όμως απορροφηθεί πλήρως μέχρι σήμερα. Τα κράτη-μέλη επίσης καθυστέρησαν στην εφαρμογή της ε, νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φύση. 20 και πλέον έτη μετά την ε, έγκριση της οδηγίας για τους οικοτόπους, πολλοί ε, τόποι και περιοχές Natura 2000 δεν έχουν ακόμα σαφή στόχους για τη διατήρηση ε, ούτε μέτρα προστασίας. Απέχουμε πόρο από την ολοκλήρωση των θαλασσίων προστατευμένων περιοχών και το θεωρώ και δικό μου έργο γιατί είμαι αρμόδιος και για την αλία και τις θαλάσσιες υποθέσεις. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις προσφυγής επί ε, παραλήψη και αυτό είναι μια δυσάριστη συνέπεια και παραμένει. Ε, άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνουν επιπλέον προσπάθειες και ενδεχομένως να αναζητηθούν νέες λύσεις. Ε, και έρχομαι τώρα στον έλεγχο της κατάστασης της φύσης. Θα ήθελα και πάλι να τονίσω ότι και ο πρώτος αντιπρόεδρος κύριος Τίμερμανς και εγώ προσωπικά τονίσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καθόλου την πρόθεση να ε, κατεβάσει το επίπεδο της ε, φιλοδοξίας για την νομοθεσία σχετικά με τη φύση. Αυτό εκφράστηκε και από πολλούς υπουργούς κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου στο, ε, το Μάιο. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι από το Refit ε, υπάρχουν πολλά προβλήματα, πολλές ευαισθησίες και ε, έχει γεννηθεί και κάποια αδημονία. Πολλοί από εσά με ρώτησαν πρόσφατα ε, τι προτιθέμεθα να κάνουμε με τις οδηγίες για τα πτηνά και για τους οικοτόπους. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι θα πρέπει να τελειώσει η δημόσια διαβούλευση και η αξιολόγηση πριν αρχίσει οποιαδήποτε συζήτηση για το τι μέλη γενέστε. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να το δούμε βεβαιασμένα χωρίς να γνωρίζουμε σε βάθος όλα τα θέματα και χωρίς να έχει γίνει απαραίτητη ε, συζήτηση και περισυλλογή. Ήδη πολύ ενδιαφερόμενοι ε, ενέχονται πάρα πολύ και αυτοί δεν είναι μόνο μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και οργανώσεις αγροτών και αλλιέων, ε, ε, ψαράδων, ερασιτεχνών και κυνηγών που ενδιαφέρονται πάρα πολύ για αυτό το εγχείρημα. Είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε να βαστούμε σε πολύ ιερά στοιχεία για να μπορέσουμε να καταλήξουμε με την πιο αποτελεσματική απόκριση και την πιο λεπτική και ευαίσθητη ταυτόχρονα αλλά και την πιο λογική. Ε, θέλω να σας πω ότι οι συνάδελφοί μου στα κράτη-μέλη υποστηρίζουν πάρα πολύ την προσέγγιση που ακολουθούμε με τις υπηρεσίες μας και ελπίζω να μπορώ να προσβλέπω και στη δική σας υποστήριξη. Η δημόσια διαβούλευση θα λήξει στις 24 Ιουλίου. Ήδη έχει ε, λάβει απαντήσεις πάνω από 200.000 και αυτή είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή ε, σε οποιαδήποτε διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι σήμερα. Τα πρώτα προκατακτικά ε, αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στις Βρυξέλλες τέλη Οκτωβρίου και ε, σας καλώ όλους να συμμετέχετε. Από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα του check-up αυτού θα κατατεθούν συνολικά στις αρχές του 2016. Τώρα, Υπάρχει και το θέμα της ενδιάμεσης αναθεώρησης της στρατηγικής βιοπικιλότητας. Η έκθεση για την κατάσταση της φύσης εγγράφεται ε, σε αυτή την προσπάθεια της ενδιάμεσης αναθεώρησης που έχει προβλεφθεί για ε, αργότερα, για το φθινόπωρο. Θα καταγραφούν η πρόοδος αλλά και οι ελλείψη στην εφαρμογή έτσι ώστε να ενημερωθούν ε, εκείνοι που παίρνουν τις αποφάσεις για το που χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει υλοποιήσει μέχρι το 2020 τις δεσμεύσεις της παγκοσμίως για την βιοπικιλότητα. Θα αποτελέσει επίσης τη βάση για τον προβληματισμό μας, για τα τομεακές ε, αναθεωρήσεις και μεταρρυθμίσεις όπως είναι η κοινή γεωργική πολιτική, αλλά και η αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αναθεώρησης επίσης θα ενημερώσουν για το πώς ε, μεταφράζονται στην πράξη οι παγκόσμιοι στόχοι για την ανάπτυξη στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα πάρα πολύ η έκθεση αυτή να είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ε, καταγραφή ή ένας προβληματισμός για το αν έχουμε φτάσει στους στόχους μας ή αν τους έχουμε χάσει θα ήθελα να είναι σε μεγαλύτερο βάθος ο έλεγχος ε, και να υπολογίσουμε το πραγματικό κόστος ε, της μη συμμόρφωσης. Ε, θα τονίσει τη σημασία της ποικιλότητας και των οικοσυστημάτων που είναι ένα πραγματικό φυσικό κεφάλαιο. Είναι κρίσιμοι τομή στους οποίους θα πρέπει να επενδύσουμε και μάλιστα πολύ σύντομα. Όπως πρόσφατα συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της πράσινης εβδομάδας, είναι σαφές ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Αυτή όμως δεν είναι αρκετή για να επιτύχουμε τους στόχους μας για το 2020. Θα χρειαστούν πολύ πιο έντονες προσπάθειες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ένταξη της βιοποικιλότητας σε διάφορες τομεακές πολιτικές και ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε με την εφαρμογή της έτσι ώστε να αξιοποιηθεί και να εκτιμηθεί αυτή η προσπάθεια και όχι να υποτιμάται όπως έχει γίνει πολύ πρόσφατα και πολύ συχνά. ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδιάζει να κάνει έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας και το καλωσορίζω πραγματικά αυτό. Χρειαζόμαστε μια νέα όθηση τώρα για να φτάσουμε στους στόχους του 2020. Μόνο εάν ενώσουμε τις τρεις διαστάσεις της αηφόρου ανάπτυξης, δηλαδή την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική πτυχή στις πολιτικές μας. Μόνο τότε λοιπόν θα είμαστε σε θέση να έχουμε μια Ευρώπη υγιή και επιτυχή που θα προσφέρει ένα μακροχρόνιο και ασφαλές μέλλον για όλους τους πολίτες της. Θα πρέπει όλοι να εργαστούμε προς μια συνολικότερη εκτίμηση της βιοπικιλότητας και των οικοσυστημάτων ως μια βάση για την υγεία και την ευημερία μας και τον πλούτο μας. Αυτό ακριβώ ήταν και το θέμα της επιτυχούς πράσινης εβδομάδας φέτος και είναι και ένα θέμα το οποίο βρίσκεται ακριβώς και στην καρδιά των θεματολογίων για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Επιτρέψτε μου τέλος να κάνω μερικά προσωπικά σχόλια. Εγώ προέρχομαι από ένα πολύ μικρό νησάκι και γνωρίζω πόσο περιορισμένες είναι οι φυσικές δυνατότητες και οι φυσικοί πόροι και τι σημασία έχει να τους φροντίζουμε για να είμαστε και οι ίδιοι ε, καλά αλλά και οι μελλοντικές γενναίες. Ε, έτσι η αρχή της ε, προφύλαξης για μένα εδώ είναι κρίσιμη. Καλύτερα να είμαστε προμηθείς παρά επιμηθείς. Η οικονομία μας, η ανάπτυξη και η θέσεις απασχόλησης θα είναι πολύ πιο διαρκής και εποφελής εάν οικοδομήσουμε ε, ε, με σεβασμό στη φύση και όχι εις βάρος της φύσης. Γι' αυτό ε, προσβλέπω σε μια ισχυρή νομοθεσία για τη φύση. Και η έκθεση για την κατάσταση της φύσης με επιβεβαίωσε σε αυτή μου την πεποίθηση. Τώρα θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα, να βελτιώσουμε την εφαρμογή, να αυξήσουμε τις επενδύσεις στη φύση και να διαχειριστούμε το Natura 2000 με καλύτερο τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας την καλοσύνη σας και περιμένω με χαρά να ακούσω τα σχόλιά σας και τις απόψεις σας. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ξεκινούμε με τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Ο κύριος Σίβο Μπέλετ από το ΕΛΚ. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε λίγο χρόνο, οπότε ένα δίλεπτο για τον κάθε ομιλήτη. Ο Ιβο Μπέλετ, ευχαριστώ. Παρά είναι σύντομο. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε στην Επιτροπή μας. Δεν θα αναφερθώ στην στρατηγική βιοπικιλότητα, στην οποία συμφώνησαν τα κράτη-μέλη και τους στόχους για το 2020 έως το 2050 μάλιστα. Θέλω να ακολουθήσουμε αυτή την άγουσα και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να, να αντιστρέψουμε αυτή την επιδείνωση των οικοσυστημάτων. Ε, διαβάσαμε πολύ προσεκτικά το χάρτη για την κατάσταση της φύσης και είπατε ότι πολλά είδη πτηνών ανακάμπτουν, αλλά ταυτόχρονα έχουμε πολλά ανησυχητικά στοιχεία που μας προβληματίζουν. Αναφερθήκατε στην ανάγκη να επενδύσουμε στη φύση. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ως προς αυτή την ανάγκη. Επίσης, ε, θα πρέπει να εναρμονίσουμε τις την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη με τη φύση. οι επενδύσεις στις ε, υποδομές δεν αφορούν μόνο το οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και άλλα θέματα που λείπουν. Ε, χαιρετίζουμε τις δημόσιες διαβουλεύσεις που θα είναι εκτεταμένες, όπως είπατε. Μας ενδιαφέρει φυσικά η έκβαση αυτών των διαβουλεύσεων και το κατά πόσο θα υποβάλλετε νέες προτάσεις σε σχέση με τις δύο πιο σημαντικές οδηγίες. Και μας ενδιαφέρει αν θα προτείνετε συνολική αναθεώρηση ή θα επικεντρωθείτε σε συγκεκριμένα άρθρα δεδομένων των σημαντικών στόχων του 2020 και του 2050. Χωρίς να είμαστε δογματικοί, αναφερθήκατε σε όλους τους ενδιαφερομένους, τους γεωργούς, τους κυνηγού, αλλά Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ε, μια συνεργασία οικολόγων και γεωργών. Δεν είναι αντίπαλοι, δεν είναι εχθροί μεταξύ τους. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν μια τέτοια συμμαχία γιατί είναι προ όφελο και των γεωργών μια φύση σε καλή κατάσταση, ένα φυσικό περιβάλλον σε καλή κατάσταση. Και χαίρομαι για τη συμμετοχή βρέω ε, φάσματο ενδιαφερομένων. Πώς θα αντιμετωπίσετε την πιθανή αναθεώρηση της οδηγίας για τα πτηνά και τους οικοτόπους. Ο Ματίας Γκρότ τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Κατά τη διάρκεια της πράσινης εβδομάδας καταδείξατε ότι το Natura 2000 είναι από τις μεγάλες ιστορίες επιτυχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι γεγονός, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αυτή η προσπάθεια, διότι από τις περιοχές ε, που έχουμε στη Natura 2000, ε, στη Χλωρίδα και την Πανίδα, στα Πτηνά, όλα αυτά είναι καλά, αλλά τα κράτη-μέλη είναι ακόμα στο στάδιο της εφαρμογής. Και τώρα μας εξέπληξε το γεγονός ότι φαίνεται ότι το Συμβούλιο θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακρούσει πρίμνα ε, και με σε αυτό που είπατε ότι δεν είναι δική σας πρόταση και πρόθεση, αλλά αυτοί που εφαρμόζουν όλα αυτά επί τόπου δεν είναι εύκολο να τα εφαρμόσουν. Στην εκλογική μου ε, περιφέρεια είχαμε μια συζήτηση για ε, την ε, οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και έγινε χαμός. Βάλανε φωτιά, κάψανε ε, διάφορα ομοιώματα, χρειαστήκαμε αστυνομική προστασία για να πάμε συνοδεία οι ευρωβουλευτές να μιλήσουμε σε μια εκδήλωση. Δηλαδή και τελικά δεν θα πρέπει να κάνουμε μια τρύπα στο νερό και να πούμε ότι το παίρνουμε πίσω και όλοι αυτοί που είναι αντίθετοι και λένε όχι σε όλα και ουρλιάζουν πιο δυνατά από όλους τους άλλους να ε, κερδίζουν. Και όπως το είπε και ο Ιβο Μπελέτ, δεν είμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον, είμαστε ο ένας μαζί με τον άλλον, γιατί το κόστος ε, έχει οφείλει και ε, είναι σαφή 5,8 εκατομμύρια ε, είναι το κόστος να εφαρμοστεί και 200 με 300 δις τελικά είναι ε, το όφελος. Μιλάνε από μόνα τους τα στοιχεία αυτά τα αριθμητικά και νομώ, νομίζω ότι θα πρέπει ε, να τα λέμε αυτά και δημόσια. Ε, δεν είναι ένα βαρύδι που κουβαλάμε, αλλά σώζουμε το περιβάλλον μας, τη ζωή μας, εκεί που ζούμε, δουλεύουμε και παράγουμε. Γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να το πούμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη συζήτηση της ε, έκθεση Δίας Πρωτοβουλίας θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, τα πούμε και να στραφούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Καλό είναι πάντα να προβληματίζεσαι αν νομοθετείς καλά, αλλά το λέω ξανά για τρίτη φορά να είναι καλή επικοινωνία για να μην καταλαβαίνει ο κόσμος ότι τα καταργείται όλα και θα πρέπει να σταματήσουν τα πάντα επί τόπου για την υπόθεση του Natura 2000. Δηλαδή αέλεγχος είναι αυτό το τσεκ που κάνετε και να μην νομίζει ο κόσμο ότι είναι ακύρωση όλων όσων έχουν γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Δεμερσμέκερ. Ευχαριστώ. Ε, ορίσατε, Επίτροπε. Σας ευχαριστώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Σας καλωσορίζω. Εγώ θα είμαι συγητής για την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Ε, κύριε Επίτροπε, πολλές φορές τα γεγονότα έχουν δίκιο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα αντιλαμβανόμαστε ε, μας προδίδει καμιά φορά. Και επειδή υπάρχει αυτή η κρίση οικονομική και χρηματοπιστωτική, ε, πολλοί κόσμος έχει την εντύπωση ότι οι οδηγίες για τη φύση ε, και για το περιβάλλον είναι εμπόδια για την οικονομική ανάπτυξη ή για τη γεωργία την ίδια. Τα γεγονότα όμως είναι εδώ. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ας πούμε, έχει καταλήξει ότι η απώλεια της βιοποικιλότητας και των οικοστημάτων είναι από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την οικονομία. Και στη δική μου την περιφέρεια, τη Φλάνδρα, έχουν γίνει εκθέσεις πολύ εύγλωτες. Οι ε, πανεπιστημιακοί στη Φλάνδρα, κύριε Επίτροπε, αυτές τις μέρες ε, ε, κρούν το θόρο, τον κόδωνα του κινδύνου στον τύπο και λένε δεν μπορούμε να φέρνουμε απέναντι την οικολογία με την οικονομία. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν για περιοχές που κοινοτομούν και αλλάζουν. Και επαναλαμβάνω, είναι θέμα αντίληψης. Ας πούμε, στο ποτάμι Σχέλντε υπάρχει ε, ένα σχέδιο που λέγεται ΣΥΓΜΑ και συμβαδίζουν οικονομική ανάπτυξη. Πηγαίνετε στην Αμβέρσα, δεν είναι μακριά, αξίζει τον κόπο να πάτε, θα δείτε εκεί και θα θαυμάσετε τι γίνεται. Για το 2015, όταν ήρθε η έκθεση για την ε, κατάσταση της φύσης, ε, όλες οι εκθέσεις λένε ότι είμαστε στο 12 παρα 5, αλλά χρειάζεται σωστά να εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα δώσει αποτελέσματα, πολλές φορές εντυπωσιακά. Και το πρώτο είναι πάρα πολύ προφανές. Δεν είναι οι οδηγίες λέει τόσο κακές, αλλά γιατί δεν εφαρμόζονται καλύτερα. Τι θα κάνουμε εμείς έτσι ώστε οι οδηγίες για τη φύση να επιβάλλονται καλύτερα, να παροτρύνονται τα κάτι μέλη, να ακολουθούν τα καλά παραδείγματα. Και αυτό το check-up θα πρέπει να βασίζεται σε γεγονότα και σε αποδείξεις. Και εγώ με μεγάλη περιέργεια γιατί με παραξένευσε αυτό που είπε ο κύριος Τίμερμανς αρχές Ιωνίου ότι η οδηγία για τα πτηνά λέει και τους οικοτόπους έχουν ξεπεραστεί και χρειάζονται ενημέρωση. Αυτό μπορεί να ισχύει αλλά γιατί προτρέχει, γιατί προεξοφλεί το αποτέλεσμα του ελέγχου. Θα πρέπει ε, κάθε μας δράση να βασίζεται σε γεγονότα, σε στοιχεία και σε αριθμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Γκερμπράντη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο που παρουσίασε την κατάσταση της φύσης στην Επιτροπή μας. Δεν πρόκειται να επαναλάβω όσα μας είπαν οι προλαλήσαντες. Εγώ θα σταθώ σε μερικά σημεία μόνο. Όπως και εσείς, ε, θα ήθελα να γνωρίσω την τεράστια επιτυχία της ισχύουσας νομοθεσίας Natura στην Ευρώπη. Αλλά το κατά πόσο εφαρμόστηκε σωστά ε, είναι συζητήσιμο, αλλά παρόλα αυτά η επιτυχία της είναι εντυπωσιακή. Πολύ σημαντικό αυτό. Η φύση μας ε, προσφέρει ό,τι χρειαζόμαστε. Η αξία της είναι ανεκτήμητη και απεριόριστη. χρήση οπωσδήποτε προστασίας ε, και διαφύλαξης. Η έκθεσή σας όμως αναφέρεται και σε κάποιες απειλές για τη φύση και τη βιοπικιλότητα και μία από αυτές είναι η γεωργία. Περίπου το 50% των, ε, της ευρωπαϊκής ε, επικράτειας είναι γεωργικές υγιές. Οπότε θα πρέπει να έχουμε στερή συνεργασία με τη γεωργική κοινότητα για να διαφυλάξουμε τη βιοπικιλότητα. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με το πρασίνισμα της κοινή μας γεωργικής πολιτικής τελικά ε, να βάγισε παταγωδός. Αλλιώθηκαν αυτές οι προτάσεις και από τα κράτη-μέλη και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αποτέλεσμα να κενωθούν περιεχομένου. Τώρα τα κράτη-μέλη ε, εφαρμόζουν και επεξεργαζόμενα τις λεπτομέρειες ε, ακυρώνουν ακόμη περισσότερο αυτή την πρόταση, την αλλοιώνουν τελείως. Τι πρόκειται να κάνετε ε, σε συνεργασία με τον Επίτροπο Φιλ Χόγκαν και τι γίνεται με τους άλλους τομείς πολιτικής, γιατί εμείς μπορούμε να επικεντρωθούμε στην νομοθεσία για τη φύση και τον μικρό αλλά επιτυχή προπολογισμό του LIFE, αλλά τι γίνεται με την πολιτική συνοχή, με την περιφερειακή πολιτική, με το επενδυτικό σχέδιο και ταμείο του Juncker. Δεν θα πρέπει να έχουμε πιο αυστηρά κριτήρια για την προστασία της φύσης και της βιοπικιλότητας και για αυτούς τους τομείς πολιτικής. Και τέλος, το οικονομικό σκέλος είναι πολύ σημαντικό, το δημοσιονομικό, γιατί γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε άπειρα κονδύλια, έχουμε 3,4 δις όμως για, την, ε, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο στο LIFE και 22 δισεκατομμύρια στο αγροπεριβαλλοντικό ε, καθεστώς. Και ε, το ελεκτικό συνέδριο διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα για το περιβάλλον, οπότε θα μπορούσαμε και εκεί και σε αυτό να επικεντρωθούμε. Τέλος, συμφωνείτε μαζί μου κύριε Επίτροπε ότι η κατάσταση της φύσης καταλήγει σε ένα συμπέρασμα, στο βασικό συμπέρασμα ότι θα πρέπει να ε, εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας όχι μόνο στην νομοθεσία της φύσης, για τη φύση αλλά και σε όλους τους άλλους, σε όλους τους άλλους τομείς. Και αν συμφωνείτε, ε, τι σκοπεύετε προκειμένου να εντατικοποιήσετε αυτές τις προσπάθειες. Ευχαριστώ κυρία Κονέτσινα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά. Παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέρον ε, αυτά που μας είπατε και περιμένω το αποτέλεσμα της διαβούλευσης. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της διαβούλευσης ε, φέρονται θετικά, αλλά ήδη έχουν περάσει δύο χρόνια και δεν έχουν γίνει και πολλά. Ελπίζω να μην ισχύσει το ίδιο και στην περίπτωση αυτή. Πάντως θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Πολύ συχνά επικρίνουμε τα κράτη-μέλη γιατί δεν στηρίζουν επαρκώς τη βιοπικιλότητα. Δεν συμμορφώνονται με τα κριτήρια, δεν μεριμνούν ιδιαίτερως για αυτήν. Αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν παραθυράκια και διαφορές. Γιατί μιλάμε για τη γεωργία τι γίνεται όμως με την υδατοκαλλιέργεια. Πόσα κονδύλια αφιερώνονται στη διατήρηση και δημιουργία υποδομών α, υδατοκαλλιέργειας, ενώ ξέρουμε τον, αντίκτυπο, τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει στη βιοπικιλότητα. Τι γίνεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τη βιομάζα. Έχουμε αντιφατικούς στόχους γιατί πολύ συχνά λέμε ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά γνωρίζουμε κάλλιστα ότι πολλές χώρες πάνε ακόμη πιο μακριά, επηρεάζοντας αρνητικά τη βιοπικιλότητα. Επίσης, πολλές φορές είναι μη αντιστρέψιμες οι βλάβες υπάρχει μια έλλειψη συνοχής και μια ασυνέπεια ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν θέλουμε να δίνουμε μαθήματα, πρώτα θα πρέπει να διορθώσουμε τα του οίκου μας. Μας είπατε επίσης ότι στα πλαίσια της στρατηγικής για τη βιοπικιλότητα και στην καταπολέμηση των χωροκατακτητικών ειδών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση τι μορφή θα λάβει αυτή η προσπάθεια περιορισμού των χώρων κατακτητικών ειδών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον Επίτροπο Βέλα που εξηγήσε τι θα κάνει και πώς θα είναι η διαδικασία. Νομίζω ότι οι περισσότερες ερωτήσεις έχουν τεθεί, για να είμαι ειλικρινής, διότι νομίζω ότι λαμβάνετε αυτή την αίσθηση εδώ της αίθουσας, ότι οι περισσότεροι δεν εμπιστεύονται αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως και μπορείτε να πείτε ότι ναι, πρέπει να εξετάσουμε τις τρέχουσες οδηγίες και κατά πόσον ε, μας δίνουν ακόμα τα αποτελέσματα που θέλουμε. Όλα ακούγονται πολύ ωραία και κανείς δεν μπορεί να είναι κατά ακούγοντάς τα. Αλλά από την άλλη υφέρπουν δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όπως είπε και ο συνάδελφος υπάρχει ο κύριος Τίμερμαντς ο οποίος ήδη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται εξυγχρονισμός. Ε, καλώς, ε, ωραία η δημόσια διαβούλευση, αλλά τι σημαίνει δημόσια διαβούλευση όταν ήδη έχει καταλήξει τα συμπεράσματά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επίσης αν δείτε τη δημόσια διαβούλευση, τονίζουμε πόσο δαπανηρή ήταν η εφαρμογή, αν οδήγησε σε θέσεις εργασίες, αν είχε κάποια προστιθέμενη αξία. Ε, Ποιο είναι ο λόγο αυτών των ερωτήσεων, όταν ο βασικό λόγο, το γνωρίζουμε όλοι, είναι η έλλειψη τη κατάλληλη εφαρμογή και δεν υπάρχει τίποτα για την εφαρμογή στη δημόσια διαβούλευση. Αυτή είναι η ουσία. Και εσείς λέτε αφενός ότι δεν θα μειώσουμε το επίπεδο της φιλοδοξίας μας, αλλά αφετέρου ρωτάτε στη δημόσια διαβίληση πόσο θα κοστίσει να την εφαρμόσουμε. Τι κάνετε ακριβώς εδώ. Πραγματικά χάθηκα λίγο σε αυτό που προσπαθείτε να, να καταφέρετε και τι ακριβώς θέλετε να προτείνετε αργότερα. Μια πολύ σαφής ερώτηση λοιπόν. Γιατί στη δημόσια διαβούλευση δεν υπάρχει καμία νήξη στην έλλειψη εφαρμογής που είναι το σοβαρότερο πρόβλημα και τι σκοπεύετε να κάνετε για να βελτιώσετε αυτό αντί να παρουσιάσετε μια οδηγία η οποία ε, ε, ξεκινήσατε και μας είπατε ότι έχει αποτελέσματα. Αν έχει αποτελέσματα και δεν θέλετε να μειώσετε το ε, επίπεδο φιλοδοξίας, ίσως θα έπρεπε να μιλάμε για την εφαρμογή της και ή την πιθανή έλλειψη εφαρμογής της και να αφήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία που μόνο έλλειψη εμπιστοσύνη δημιουργεί. Ευχαριστώ κύριο Σπιντιτσίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Εγώ θα συνεχίσω από τα όσα είπε ο Μπάς Αικχάουτ και θα κάνω μια πολύ σύντομη ερώτηση. Η έκθεση της ε, κατάστασης της φύσης μας δείχνει ότι η βιοποκυλότητα στην Ευρώπη επιδεινώθηκε περαιτέρω τα τελευταία χρόνια και υπάρχουν όμως και κάποιες επιτυχημένες ιστορίες όπου οι οδηγίες για τη φύση εφαρμόστηκαν πλήρως με πάσα λεπτομέρεια και ως αποτέλεσμα κάποια είδη ε, επανήλθαν στην αρχική τους κατάσταση, για παράδειγμα οι κάστορες ε, και διάφορα άλλα ζώα. Για να συνεχίσω λοιπόν από την ερώτηση του Μπέας Άικχο. Τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώπιον των κρατών μελών που αντίθετα με αυτά που σας ανέφερα δεν εφαρμόζουν σωστά τις οδηγίες και έτσι δεν επιτρέπουν στους πολίτες να απολαμβάνουν ε, των ωφελών τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο για να δώσετε τις απαντήσεις σας, τις οποίες περιμένουν οι συνάδελφοι. Καταρχάς σας ευχαριστώ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και θα ήθελα να ξεκινήσω με τον Ιβο Μπέλετ. Όσον αφορά την πρόοδο για την κατάσταση της φύσης. Να είμαι σαφής. Στην αρχή είχαμε την έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος, μετά είχαμε την έκθεση για την κατάσταση της φύσης, η οποία επιβεβαίωσε αυτά τα οποία είχαμε ήδη ε, πει ότι όντως έχει υπάρξει κάποια πρόοδος, αλλά παρά το γεγονός ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος, δεν έχουν ε, επιτευχθεί όλοι οι στόχοι. Και πέραν αυτού και οι δύο εκθέσεις κρούν τον γόνατο του κυρδίνου. Ότι στο μέλλον, εάν συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που κάναμε, τότε τα πράγματα θα επιδεινωθούν, τα προβλήματα θα επιδεινωθούν. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι εξή. Μετά από την έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος, μετά από την έκθεση για την κατάσταση της φύσης, θα αφήσουμε τα πράγματα να κυλήσουν ως έχουν. Και αυτή η ερώτηση δεν απαντάτε μόνο από μένα, δεν αποφασίζω μόνο εγώ, είμαστε όλοι συνένοχοι και θα πρέπει να το συζητήσουμε και να βρούμε μια λύση από κοινού. Όσον αφορά τη δημόσια διαβούλευση, θεωρώ ότι οι στόχοι θα παραμείνουν πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας. Ήβο, αναφέρθηκε επίσης και στους γεωργούς και θα επανέλθω στο θέμα αυτό, διότι είπε ότι οι γεωργοί είναι η σύμμαχοί μας και η καλύτερη μας φίλη. Θα ήθελα να επαυξήσω εδώ, διότι Θέλω να πω ότι η καλή γεωργία είναι η συμμαχή μας, η καλή γεωργία είναι η φίλη μας, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όπως υπάρχει καλή γεωργία και καλή καλλιέργεια, υπάρχει και κακή γεωργία και κακή καλλιέργεια. Και επομένως θα πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό. Ματίας, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σου. Για το Natura 2000, πράγματι έχει υπάρξει πρόοδος, ιδίως όσον αφορά τη γη, τις γης, αλλά Όταν γίνεται λόγος για βιοπικιλότητα, σχεδόν πάντα λησμονούμε ότι έχουμε βιοπικιλότητα ε, στο 30% του πλανήτη και έχουμε και βιοπικιλότητα στο υπόλοιπο 70% του πλανήτη, δηλαδή τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας. Στην ξηρά έχουμε το 17% των εκτάσεων μας στο Natura 2000 και στις θάλασσες και στο ωκεανούς έχουμε μόνο 4%. Συμφωνώ απολύτως με τον Ματίας ως προς το γεγονός ότι δεν θα πρέπει ε, να υπαναχωρήσουμε ε, σε αυτό τον έλεγχο της κατάστασης. Δεν πρέπει και δεν μπορούμε να υπαναχωρήσουμε, αλλά θα πρέπει να έχουμε το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Κάποιες φορές υποπίπτουν σε εξή σφάλμα. Κοιτάμε να δούμε κατά πόσο οδηγία μπορεί να καλύψει τις σημερινές προκλήσεις. Οι σημερινοί στόχοι μπορεί να καλύψουν τις σημερινές προκλήσεις. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι προκλήσεις του μέλλοντος είναι πολύ μεγαλύτερες από τις σημερινές και πρέπει να σκεφτόμαστε με βάση το μέλλον και να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με βάση το σήμερα. Πρέπει να σκεφτούμε τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Αυτά είναι προγράμματα και στόχοι τα οποία θα μπορούν σου να μας βοηθήσουν να έχουμε επιτυχίες. Ξέρω ότι ο Ματίας είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία στην περιφέρειά του για το πρόγραμμα αυτό με τα ύδατα Τι γίνεται λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έχουμε κάποιες επιτυχημένες περιπτώσεις ε, και εξετάζουμε το κόστος και την ωφέλεια. Ναι, μένουν καλά, αλλά δεν αρκούν. Πολύ συχνά όταν εξετάζεται το κόστος, η σχέση κόστος-οφελίας εξετάζεται μόνο με βάση χρήματα. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι δώσαμε 100 και πήραμε όφελος 80 πολύ σπάνια ε, προσθέτουμε στην εξόρισωση και τα περιβαλλοντικά ωφέλη. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ξανασκεφτούμε τα πράγματα. Ο κύριος Ντέμες Μάκερ, ο οποίος θα είναι και ο εισηγητής, και χαίρομαι που θα συνεργαστούμε επί του ζητήματος αυτό. Η αντίληψη που έχουμε για τις οικονομικές πιέσεις Δυστυχώς υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι το περιβάλλον αποτελεί πάντα πρόσκομα στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά ευτυχώς αυτή η αντίληψη, αυτή η νοοτροπία αρχίζει να αλλάζει και επομένως θα πρέπει να δώσουμε και εμείς μια μάχη για να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Σήμερα πολλοί, ε, ιδιαίτερα η νέα γενιά, αντιλαμβάνονται ότι η οικονομία μας εξαρτάται από τη βιοπικιλότητά μας. Σκεφτείτε οποιοδήποτε προϊόν οποιοδήποτε κατασκευασμένο προϊόν. Μπορούμε να ε, βρούμε ποια ήταν η πρώτη ύλη από τη φύση, από τη βιοποικιλότητα. Επομένως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Εάν δεν φροντίσουμε εμείς τη βιοποικιλότητά μας, δεν φροντίζουμε και την οικονομία μας. Και απόδειξη αυτού είναι και το γεγονός ότι ακόμα και στη διάρκεια της κρίσης, ο καλύτερος τομέα, τομέας, αυτός ο οποίος συνέχισε να αναπτύσσεται, ήταν ο τομέας της πράσινης ανάπτυξης, των πράσινων θέσεων εργασίας, εν καιρό κρίσης. Επομένως, η άποψη ότι το περιβάλλον αποτελεί πρόσκομα είναι καθόλου λανθασμένη. Και δεν νομίζω ότι είμαστε μόνο εμείς. Εμείς είμαστε οι νομοθέτες. Συζητούμε, ε, νομοθετούμε, ε, φροντίζουμε να εφαρμόζονται οι νόμοι, αλλά ο ιδιωτικός τομέας το αντιλαμβάνεται αυτό και όταν ο ιδιωτικό τομέα αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να φροντίσουμε τη βιοπικιλότητα, τότε αρχίζει να επενδύει. Και ο ιδιωτικό τομέα έχει ήδη αρχίσει να επενδύει σε μία σειρά από ε, πράσινους τομείς, στην κυκλική οικονομία και ούτω καθεξής. Όσον αφορά το θέμα της εφαρμογής, συμφωνώ απολύτως, η εφαρμογή πάντα είναι το σημείο στο οποίο θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Κύριε Γκερμπράντι, πράγματι η ισχύησα νομοθεσία έχει επιφέρει κάποια αποτελέσματα, αλλά, επαναλαμβάνω, δεν μας δίνει όλα τα αποτελέσματα και δεν επιτυγχάνουμε όλους τους στόχους μας. Ε, πρέπει πριν αρχίσουμε να εξετάζουμε οτιδήποτε άλλο, να εξετάσουμε και το θέμα της εφαρμογής. Η φύση είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή μας, είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Εξαρτώμαστε απολύτως από τη φύση και όπως είπατε κι εσείς, η φύση μας προσφέρει πάμπολες υπηρεσίες χωρίς ποτέ να μας στέλνει το λογαριασμό. Και πολύ συχνά λέω ότι χρειαζόμαστε τη φύση περισσότερο από ότι η φύση χρειάζεται μας. Εάν φερθούμε καλά στη φύση, η φύση θα μας φερθεί καλύτερα. Αν φερθούμε άσχημα στη φύση, τότε η φύση θα μας φερθεί χειρότερα. Όσον αφορά τη γεωργία, συμφωνώ μαζί σας. πρέπει να κάνουμε διαφοροποίηση μεταξύ καλής και κακής γεωργίας, καλής και κακής καλλιέργειας. Ε, σύντομα θα έχουμε την αναθεώρηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ε, στην κοινή γεωργική πολιτική έχουμε 30% των κονδυλίων που θα έπρεπε ε, να είναι αφιερωμένα στο greening, στο μετριασμό των επιπτώσεων ε, του, στο περιβάλλον. Και επομένως θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα κονδύλια αυτά στην κοινή γεωργική πολιτική. Όσον αφορά τη γεωργία, προς το παρόν η άποψη δική μου είναι ότι εάν δεν επιδοτούμε επιζήμιες ε, ουσίες ε, για την ενέργεια, τότε βάσει του ίδιου επιχειρήματος, αν έχουμε επιζήμιες ουσίες και για τη γεωργία, θα πρέπει να σταματήσουμε να τα επιδοτούμε. Εάν η κακή γεωργία είναι εις βάρος των υδάτων μας, των εδαφών μας, ε, του αέρα μας, τότε σκοτώνει την ίδια τη γεωργία που εξαρτάται από αυτά. για τη συνεργασία με τον συνάδελφό μου, τον Φιλ Χόγκαν. Έχουμε ήδη ξεκινήσει συζητήσεις και αν χρειαστεί θα αναλάβουμε δράση από κοινού. Ναι, συμφωνώ και εγώ ότι η έκθεση για την κατάσταση της φύσης λέει ότι θα πρέπει να ε, αυξήσουμε τις προσπάθειές μου και όταν με ρωτούν τι θα κάνω εγώ, ε, απαντώ ότι δεν έχει σημασία τι σκοπεύω να κάνω εγώ, πρέπει να κάνουμε κάτι από κοινού. Το εμείς είναι αυτό το οποίο έχει σημασία εδώ. Τώρα, τι θα κάνουμε με τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης. Νομίζω ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική διαδικασία. Εμείς δεν θα αποφασίσουμε τίποτα, προτού λάβουμε υπόψη όλες τις ε, ε, απαντήσει τα σχόλια, τις ιδέες που θα προκύψουν από τη δημόσια διαβούλευση. Όντως κάποια κράτη-μέλη επικρίνονται συνεχώς ότι δεν ε, ε, υποστηρίζουν τη βιοπικιλότητα και θα πρέπει εκεί να συνεχίσει η εφαρμογή, να συνεχίσει η παρακολούθηση. Όσον αφορά την έλλειψη συνέπειας στην νομοθεσία, νομίζω ότι η νομοθεσία είναι ίδια. Η συνέπεια είναι στον τρόπο εφαρμογής. Υπάρχουν 28 κράτη-μέλη τα οποία ε, τρέχουν με 28 διαφορετικές ταχύτητες. Αν θέλουμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι, θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι ως προς τα αποτελέσματα, θα πρέπει να βρούμε ποια κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία υστερούν, να δούμε γιατί υστερούν και αν και εφόσον χρειαστεί θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τα υποστηρίξουμε. Λοιπόν, εξετάζουμε και το θέμα των χωροκατακτητικών ειδών, εξετάζουμε τις αρνητικές συνέπειες ε, φαινομένων που εμφανίστηκαν πριν από 10, 15, 20 χρόνια τα χωροκατακτητικά είδη ε, δεν θα μας δείξουν ε, τις αρνητικές του συνέπειες αμέσως, αλλά πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι αυτές οι συνέπειες θα φανούν στο μέλλον. Κύριε Εκχάουτ. Το γεγονός ότι ε, οι πολίτες δεν εμπιστεύονται αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο δεν μας επιτρέπει να συνεργαστούμε και να προχωρήσουμε μαζί είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης. Πρέπει να αρχίσουμε να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον και να μιλήσουμε ειλικρινά. Είπατε ότι ίσως ε, οι πολίτες δεν εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω το ίδιο. Εμπιστεύεστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγγυηθεί ότι δεν θα οπισθοδρομήσουμε εάν για παράδειγμα ε, αλλάξουμε την οδηγία για τα πτηνά. Ε, πρέπει να αρχίσουμε να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Εάν λοιπόν δεν εμπιστεύεστε εσείς τους συνάδελφούς σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να το πείτε. Μην αρχίσετε να κατηγορείτε τον Τζοβάνι, εμένα ε, ή οποιονδήποτε άλλο. Ε, να μιλάμε ειλικρινά και να ανοίξουμε τα χαρτιά μας. Ναι, ο κύριος Ντίμερμαν σας έδωσε μια εγγύηση, εγώ σας εγγυώμαι, αλλά αν υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης, τότε δεν θα υπάρξει καμία δράση εάν δεν υπάρξει συνένεση για αυτή τη δράση. Και αναφερθήκαμε και στην έλλειψη εφαρμογής και το κόστος της εφαρμογής. Εγώ δεν αναφέρομαι στο κόστος της εφαρμογής, αναφέρομαι στο κόστος της μη εφαρμογής της νομοθεσίας, διότι το κόστος της μη εφαρμογής της νομοθεσίας είναι πολύ μεγαλύτερο. Το επιχείρημά μου λοιπόν είναι μη μου πείτε πόσο στοιχίζει η εφαρμογή, πείτε μου πόσο στοιχίζει η έλλειψη εφαρμογής. Διότι αν ε, δεν εφαρμόσουμε κάτι, το κόστος είναι πάντα πολύ ψηλότερο. Ναι, η νομοθεσία που έχουμε έχει αποτελέσματα, οι πολιτικές μας επιφέρουν αποτελέσματα, αλλά και πάλι εξετάζοντας την έκθεση για το περιβάλλον, την έκθεση για τη φύση ε, και επειδή υπάρχει ενδιάμεση αναθεώρηση, ο καθένας από εμά θα πρέπει να δει τα πράγματα, να πει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, υπήρξε πρόοδος, δεν φτάνει αυτή η πρόοδος, εάν να δρανίσουμε τότε θα έχουμε περισσότερα προβλήματα στο μέλλον. Εάν αφού εξετάσουμε αυτές τις εκθέσεις, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε τίποτα, όπως σας είπα δεν επαφίεται μόνο σε μένα, επαφίεται σε όλους μας να δράσουμε. Και τέλος, ε, νομίζω ότι απάντησα ε, στο ερώτημα του κυρίου Πιεντιτσίνη για τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης και τη σημασία της και τη σημασία όχι μόνο της ευρωπαϊκής φύσης, διότι όταν αναφερόμαστε στη βιοποικιλότητα δεν μπορούμε απλώς ε, να περιοριστούμε στα ευρωπαϊκά ε, όρια. Δεν μπορούμε σήμερα να αναφερόμαστε σε ευρωπαϊκή βιοποικιλότητα ή κινέζικη βιοποικιλότητα ή αμερικανική βιοποικιλότητα. η κινεζικη βιοποικιλοτητα η αμερικανικη βιοποικιλοτητα ένα περιβάλλον για κάθε χώρα. Σήμερα είναι παγκόσμια τα θέματα, είναι παγκόσμιο το περιβάλλον και πρέπει να υπάρξουν παγκόσμιες λύσεις. Γι' αυτό και ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δεσμευτεί περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Επίτροπε. Και τώρα θα ξεκινήσουμε το δεύτερο γύρο. Έχουμε εννέα συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο. Αλλά δυστυχώς έχουμε μόνο 20 λεπτά στη διάθεσή μας. Γι' αυτό παρακαλώ υποβάλλετε τις ερωτήσεις σε ένα λεπτό. Θα τις συγκεντρώσουμε και θα τις ε, απαντήσει ομαδικά ο Επίτροπος Ιάννη Συριαπήρικ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω στον Επίτροπο ότι θέλω να το, μπορώ να τον εμπιστεύομαι. Αλλά το 2007 είχα δει στην Ολλανδία ότι είχαμε 62 ε, ε, τομείς ε, Natura 2000 με χίλια είδη χλωρίδας και πανίδας. Εκεί οι αγρότες εδώ και αιώνες ζουν σε αυτά τα μέρη και τώρα δεν μπορούν ε, να πάρουν άδεια για νέους στάβλους γιατί υπάρχει το πρόβλημα με την αμμονία και με τα αζωτούχα και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μα πρόκειται για οικονομική, κοινωνική ε, και περιβαλλοντική πτυχή. Στη χώρα μου λέει ο δικαστής που τα εφαρμόζει όλα αυτά, ε, γιατί το δίκαιο είναι σημαντικό και ο δικαστής τα ορίζει αυτά και είναι κρίμα και θα πρέπει να κλείνουν τώρα γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Μα πώς γίνεται αυτό. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν στη στάση μας ε, συνεπής με μέτρο. Ελάτε σας παρακαλώ στη περιφέρειά μου να δείτε ανθρώπους καλούς, εργαζόμενους, αγρότες που θέλουν να συνεργαστούν και βγαίνει ο δικαστής και σου λέει το απαγορεύει η Ευρώπη αυτό. Και ε, πρέπει να σας πω ας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς. Ευχαριστώ πολύ κύριο Ντάνς. Um, ευχαριστώ και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Υπάρχει μεγάλη διαφορά το πώς αντιλαμβανόμαστε τον αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και στην πραγματικότητα. Πολλοί κλάδι ε, και στα ορυχεία και αλλού είναι υπέρ της οδηγίας για τους βιότοπους, γιατί η σωστή εφαρμογή της εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου και συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού. Τι μπορείτε να κάνετε και εσείς αλλά και εμείς, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να γεφυρωθεί αυτή, αυτό το χάσμα μεταξύ ε, παρεξηγημένης αντίληψης, ε, παρανόησης και πραγματικότητας, γιατί αυτό υπονομεύει την πρόοδο μας, αυτή η παρεξήγηση. Ευχαριστώ, κύριε Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ. Α, θέλω να ρωτήσω για τη Γεωργία. Πολλά ακούσαμε σήμερα από τους συναδέλφους από την Επιτροπή Γεωργίας. Είναι σαφές ότι η Ευρώπη δεν παράγει αρκετά τρόφιμα δεν έχουμε αυτάρκεια. Η πατρίδα μου ούτε τα μισά προϊόντα που χρειαζόμαστε για κατανάλωση δεν παράγουμε. Έχουμε ένα πρόβλημα λοιπόν εκεί. Τι γίνεται σε επίπεδο υψηλό στρατηγικού σχεδιασμού. Γιατί αν στηρίξουμε αυτή την έκθεση για την κατάσταση της φύσης, τότε από πού θα εξασφαλίζουμε τα τρόφιμά μας και αν εφαρμόσουμε μέτρα πρασινίσματος. Τα, πιο βαριά απέτυχαν. Μα τώρα μόλις άρχισαν να εφαρμόζονται. Τα υπόλοιπα θα λειτουργήσουν σωστά είναι υπεραπλουστευμένα, υπεραπλοϊκά. Γιατί θέλουμε υψηλότερη παραγωγικότητα και μεγαλύτερη, ε, πιο αποτελεσματική για να, και να αφήσουμε παρόλα αυτά ένα ε, χώρο για τη φύση ή θα χρειαστεί να εισάγουμε μαζικά αυτά που πρέπει να καταναλώσουμε. Ευχαριστώ κύριο Σφαρία. Ευχαριστώ. Αγαπητέ Επίτροπε, όπως συνέβη και με τους στόχους του 2010, τα στοιχεία μας δείχνουν ότι εξαιτία πολλών παραγόντων δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε την απώλεια βιοπικιλότητας μέχρι το 2020. Κάθε χρόνο χάνουμε το 3% του ΑΕΠ εξαιτία τη απώλειας βιοπικιλότητας. Παρά τα σημαντικά νομοθετικά μέτρα που έχουν θεσπιστεί ε, προκειμένου να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι, όπως η οδηγία για τα πτηνά και τα ενδιατήματα, για το είδωρο, για τη στρατηγική για τη θάλασσα, η κοινή γεωρική πολιτική και η κοινή αλληλευτική πολιτική. Είναι ε, λογική είναι γνωστές οι συνέπειες της ε, η η εντατική γεωργία, η υπερβολική εντατική γεωργία, δασοκομεία, ε, μόλυνση, χωροκατακτητικά είδη, ε, μερικές φορές και η αστική ανάπτυξη, συμβάλλουν όλα αυτά στην απώλεια βιοπικιλότητας. Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Χρειαζόμαστε περισσότερη κοινοτική νομοθεσία ή να συμπεριλάβουμε περισσότερα θέματα βιοποικιλότητας σε άλλους κλάδους όπως Γεωργία και Ελία ή είναι θέμα ε, κακή συμμόρφωση σε κρατικό επίπεδο και πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ κύριος Εκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε Βέλα που μπήκατε στον κόπο να έρθετε στην Επιτροπή μας για να έχετε μια ανταλλαγή απόψεων μαζί μας. Χάρηκα ιδιαίτερα από αυτό που είπατε για τους φιλόδοξους στόχους που έχετε, τους οποίους και μας παρουσιάσατε. Και ακούγοντάς σας, τουλάχιστον εγώ σας εμπιστεύομαι. Και μ' αρέσει αυτό που λέτε για καλούς και κακούς αγρότες. Διότι ποιος οδήγησε ιδιαίτερα στο να υποχωρεί η βιοπικιλότητα. Από τη μια ήταν οι αγρότες και στους ωκεανούς ήταν οι αλείς που έχουν αδειάσει τους ωκεανούς από τα ψάρια. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή απέναντι σε αυτές τις κατηγορίες. Εκτός αν έχουν κάνει οι αγρότες ένα άλμα εξελικτικό που θέλουν την ευημερία τους να είναι εις βάρος ε, της ευημερίας της φύσης και των υπολείπων ειδών. Τα ίδια και στην αλία ισχύουν. Και ρωτώ, τώρα εσείς επιδιώκετε κάποιους στόχους. Ε, κανένα χρονοδιάγραμμα θα μας φέρετε και πότε μπορούμε να υπολογίζουμε σε αυτό. Thank you very much. And now, Mr. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σε ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε. Κάνετε πολλέ δηλώσει για το τι σκοπεύετε να κάνετε. Αυτό που διαβάζω εγώ στην έκθεση για τη φύση θέλουμε να δούμε κάτι για τη βιοπικιλότητα, εκεί ακριβώς οι οδηγίες για τη φύση εφαρμόστηκαν καταλήλως. Αυτό δεν είναι κάτι που το λέω εγώ. Οι συντονιστές ε, της Ευρωπαίας ε, της Επιτροπής ε, συμφώνησαν ότι δεν χρειάζεται να αναθεωρηθεί η οδηγία Natura. Ε, ε, πώς κατέληξε στο συμπέρασμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειαζόμαστε να κάνουμε μια αναθεώρηση της οδηγίας. Μήπως ο κύριος Γιούνκερ ξύπνησε ένα πρωί και είπε ότι θεωρεί ότι χρειαζόμαστε μια αναθεώρηση. Δεύτερον, είπατε ότι ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να αντιληφθεί ότι η πράσινη οικονομία είναι το μέλλον. Ε, νομίζω όμως ότι είναι πολύ περίεργος τρόπος να προσπαθούμε να τους πείσουμε για κάτι τέτοιο, ξεκινώντας μια αναθεώρηση της οδηγίας Natura. Επίσης θεωρώ ότι αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα είναι να ανοίγει το κουτί της Πανδώρας. Ε, όλοι μπορούμε να φανταστούμε ποιο είναι το επίπεδο των ε, ε, πιέσεων από τα λόμπι και το τι ακριβώς θα γίνει με την οδηγία για το Natura τους επόμενες μήνες και θεωρώ ότι έχουμε μπει σε πολύ επικίνδυνα νερά. Χωρίς μικρόφωνος ο πρόεδρος, η κυρία Έμι. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε, ευχαριστώ που απαντάτε στις ερωτήσεις μας. Εγώ θα συμφωνήσω με τις απορίες των συναδέλφων που έχουν προκύψει όλοι, ε, από όλους από την έκθεση για την κατάσταση της φύσης. Βλέπουμε ότι οι δείκτες επιδεινώνονται. Το 70% των κοινοτικών φυσικών οικοτόπων ε, είναι κάτω από τις προδιαγραφές που έχει καθαρίσει η οδηγία Habitat και ε, το 70% των ειδών ε, αντίστοιχα βρίσκονται κάτω από τα πρότυπα τα οποία θα πρέπει να τηρούνται. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μήπως θεωρείτε ότι και οι ε, πολιτικές που σχετίζονται με την ε, χρήση της γης ε, και με τη χρήση τσιμέντου και τη, που αφορούν τις αστικές περιοχές ε, θα υποσκάψουν τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή και μάλιστα με πολύ ευαίσθητα τρόπο και σε σχέση με τις πολύ λίγες καλές περιπτώσεις που γνωρίζουμε. Θα πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη και ότι όλες οι δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να ε, την χάνουν και αντίστοιχων κινήτρων και έχουν πολύ σημαντικές και οικονομικές επιπτώσεις. Και μία τελευταία ερώτηση. Ο αριθμός των παραβιάσεων οι διαδικασίε επί παραβάση που είναι εκρεμείς αυτή τη στιγμή και να σας υπενθυμίσω και πόσε αναφορές λαμβάνουμε στην Επιτροπή Αναφορών που αποτελούν ένδειξη του ενδιαφέροντος των πολιτών για τα θέματα αυτά. Ε, θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Colin Η κυρία Κόνι Λάγκεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε Βέλε, η νομοθεσία για τη φύση, για τα πτηνά και τα λοιπά, αυτό το καιρό εξετάζονται. Ε, κατά πόσο η νομοθεσία είναι επίκαιρη και ε, ε, αυτό με βρίσκει σύμφωνη. Η REFIT σημαίνει να είναι λιγότερο γραφειοκρατικές οι οδηγίες, πιο ε, καλύτερες και εύκολες στην εφαρμογή τους και εγώ είμαι η πρώτη που θα το προσυπογράψω. Αλλά δεν θα πρέπει αυτό να χρησιμοποιηθεί ως πρόφαση ε, έτσι ώστε από το παραθυράκι να καταργηθεί η νομοθεσία ή να μειωθεί η προστασία. Πολλές φορές ε, φταίει η κακή εφαρμογή στα κράτη-μέλη και στην προστασία της φύσης υπάρχει πολύ μεγάλο έλλειμμα που πρέπει να καλυφθεί διότι πολύ πόμεθα. πολύ. Εσείς ως Επίτροπος πώς θα εξασφαλίσετε ότι δεν θα αποδυναμωθεί η ε, νομοθεσία με την πρόφαση της άρσης της γραφειοκρατίας. Ευχαριστώ κυρία Μέλια. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο Βέλα. Εγώ είμαι αγρότησα. Ε, είναι ένας κλάδος όπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα και θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα καταφέρουμε το πρασίνισμα αυτό να αξιοποιηθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βιολογική ποικιλότητα. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Μέχρι τώρα υπάρχει η 15η Μαΐου που είναι μια προθεσμία ε, για ε, την αμυψισπορά ε, για γέες που βγαίνουν από την αγρανάπαυση και αλλάζουν χρήση και καλλιέργεια. Εγώ το έχω δει και στην ίδια μου τη γη πώς καταστρέφεται μια προσπάθεια ε, ε, που έχουμε κάνει χρόνια ολόκληρη. Αν αλλάξει λίγο αυτή η ημερομηνία θα ξανά έχουμε τα οδικά πτηνά και διάφορα αποδημητικά ε, ξανά στα χωράφια μας. Δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να φύγει ο Επίτροπος. Θα του δώσω αμέσως το λόγο να απαντήσει όσο μπορεί ομαδικά. A Ευχαριστώ. Λίγα σύντομα σχόλια. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια του συναδέλφου από την, συναδέλφου από την Ολλανδία. Συμφωνώ, όπως είπα και προηγουμένως. Δεν μπορούμε όμως να λέμε ότι όλες οι ιερικές δραστηριότητες είναι καλές ή κακές και να γενικεύουμε, να τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Το ίδιο ισχύει και για την Ελία. Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτή η γενίκευση. Καθήκον μας είναι να διαφοροποιούμε, να ψάξουμε τους καλούς και να τους διαχωρίσουμε από τους κακούς και κάποιος θα πρέπει να υπομειστεί την ευθύνη. Κύριε Ντάνς, σε ό,τι αφορά την ανισορροπία και τη διαφορά μεταξύ ε, της αντίληψης, της φαλμένης αντίληψης και της πραγματικότητας. Ναι, οι εκθέσεις αυτές μιλούν για την κατάσταση του περιβάλλοντος, για την κατάσταση της φύσης και κατά τη γνώμη μου αυτές οι εκθέσεις είναι το μόνο εργαλείο που μπορεί να διαλύσει τις παρεξηγήσεις, ε, τις ασφαλμένες αντιλήψεις. Και όταν συζητούμε τις πολιτικές θα πρέπει να λάβουμε αποφάσεις για δράσεις με βάση αυτές τις ε, τεκμηριωμένες εκθέσεις και όχι με βάση κάποιες αντιλήψεις ή κάποιες ιδέες. Συμφωνώ πάντως ότι πρέπει να κάνουμε διαφοροποίηση μεταξύ αντίληψης και πραγματικότητας. Κυρία Γκέρλινγκ, ναι, και πάλι το γεωργικό ζήτημα ανέκυψε. Ακόμη και εδώ όμως ε, θεωρώ ότι δεν υπάρχει άλλος τομέας που μπορεί να βρει λύσεις, γεωργικές λύσεις για καλύτερη γεωργία παρά μόνο ο ίδιος ο κλάδος της γεωργίας. Και συμφωνώ μαζί σας ότι δεν παράγουμε αρκετά τρόφιμα, αλλά έχουμε επιλογές. Σήμερα είναι γεγονός ότι 80% των τροφίμων μας το βγάζουμε από το 30% του πλανήτη μας. Το λέω και το επαναλαμβάνω και δεν θα κουράζομαι να το λέω. Είτε μας αρέσει είτε όχι πρέπει να στραφούμε προς τους ωκεανούς. Μπορεί να διαφωνείτε, αλλά ο αυτός ο αιώνας, ο αιώνας μας θα πρέπει να είναι ο γαλάζιος αιώνας. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να παρατραβούμε και να υπερεκμεταλλευόμαστε μία ε, ε, οικονομία που στηρίζεται στην ξηρά. Ε, σε 7 δισεκατομμύρια τώρα, μετά θα χρειαστούν πολύ περισσότερα. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε παόριστο χωρίς να πιέζουμε τη βιοπικιλότητα. Πρέπει να στραφούμε από την ξηρά στη θάλασσα. Πριν από λίγες μέρες ξεκινήσαμε διεθνείς δημόσιες διαβουλεύσεις για την καλύτερη διακυβέρνηση των θαλασσών και ωκεανών. Γιατί πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας προς τον ωκεανό και για την ενέργεια, για να βρούμε εναλλακτικέ πηγές ενέργειας, για να βρούμε εναλλακτικά ε, πηγές τροφίμων, για εναλλακτικές ε, επιλογές στην οικονομική ανάπτυξη και εκεί θα πρέπει να αναλάβετε το ρόλο σας κι εσείς, γιατί θέλουμε να στραφούμε προς τους ωκεανούς για τις οικονομικές δυνατότητες που δίνουν και θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο και για τις περιβαλλοντικές ευθύνες που υπάρχουν. Γι' αυτό και θα πρέπει στο μέλλον να συζητήσουμε τις περιβαλλοντικές ευθύνες που θα πρέπει να αναλυφθούν όταν μιλούμε για τους ωκεανούς μας. Σήμερα βέβαια δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την οικονομία ή τη γεωργία ή την αλληλεία. Σήμερα θα πρέπει να, μιλήσουμε, να μιλούμε για αηφόρο οικονομία, για βιώσιμη γεωργία, για βιώσιμη αλία, για αηφόρο τουρισμό. Οτιδήποτε δεν είναι βιώσιμο έχει ημερομηνία λήξης. Έτσι πρέπει να δράσουμε. Δεν θέλουμε μια απλή γεωργία. Θέλουμε βιώσιμη γεωργία. Δεν θέλουμε ε, απλώς μια αλία. Θέλουμε βιώσιμη αλία. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο αν δεν είναι βιώσιμο. Σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις της βιοπικιλότητας. Οι εκθέσεις ε, ε, επισημαίνουν την πρόκληση της εφα... σωστής εφαρμογής. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι πάντα πρόκληση η εφαρμογή. Όταν όμως η έκθεση ε, επισημαίνει μια σειρά πιέσεων απειλών και προκλήσεων στη βιοπικιλότητά μας, οι τρεις βασικές προκλήσεις, η πρώτη είναι η γεωργία. Η γεωργία από μόνη της αντιπροσωπεί το αντιπροσωπεύει το 25% της πίεσης ε, στην ε, βιοπικιλότητα. Και οι τρεις πρώτες πιέσεις είναι πάνω από το 50% της συνολικής πίεσης προς την ε, βιοπικιλότητα. Αν λοιπόν μιλούμε για πιέσεις που ίσως δεν ελήφθησαν υπόψη στο παρελθόν, θα πρέπει να συνεχιστούν να μελούνται και σήμερα Κύριε Εκ, για το χρονικό πλαίσιο. Ο χρονικός ορίζοντας ε, είναι το 2020, οπότε όλοι μας οι στόχοι έχουν ένα χρονοδιάγραμμα και αυτό λύγει το 2020. Το 2020 πρέπει να υλοποιήσουμε τους στόχους ήδη, όχι να ξεκινήσουμε τη δράση το 2020. Σε ορισμένου τομεί ήδη στερούμε και έχουμε καθυστερήσει στην ανάληψη δράσεων. Οπότε το χρονικό πλαίσιο είναι τώρα. Η προθεσμία για την υλοποίηση των στόχων το αργότερο το 2020. Για την υλοποίηση όμως. Κύριε Γιάμπορ. Ναι. Οδηγίες για τη φύση. Ναι, αποδίδουν καρπούς όπως είπα οι οδηγίες για τη φύση. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνομαι. Ο έλεγχος καταλληλότητας, το fitness check, δεν σημαίνει αναθεώρηση μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων μπορεί να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα. Αλλά διαβούλευση χρειάζεται για να διαπιστώσουμε κατά πόσο χρειάζεται κάποια αναθεώρηση ή όχι. Όπως είπα, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα απολύτως αν δεν λάβουμε υπόψη τις παρατηρήσεις ε, και ε, τα αποτελέσματα της ε, διαβούλευσης. Για τις πολιτικές για τη γη, ε, μη βιώσιμες αποφάσεις για τη γη ήταν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη βιοπικιλότητά μας αρνητικά. Φυσικά θα πρέπει να προσέξουμε τη χρήση της γης. Για την εφαρμογή θα πρέπει όλα τα κρατημέλη να εφαρμόσουν τις οδηγίες, να μειώσουν τη γραφειοκρατία και συμφωνώ. Οι στόχοι είναι και υπάρχουν, θα πρέπει να παραμείνουν, ίσως και να ενισχυθούν. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως να βρούμε ε, ευφιέστερους τρόπους για να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους. Και αυτή είναι η έκκλησή μου. Σας παρακαλώ, σας θέρμα παρακαλώ να συνεργαστούμε για τα θέματα αυτά. Σήμερα το πρωί είδα ότι ήταν πολύ ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την κυκλική οικονομία. Διαπίστωσα ότι το Κοινοβούλιο στηρίζει σύσσωμο τον κοινό αυτό στόχο της κυκλικής οικονομίας και με χαροποιεί ιδιαίτερα σε αυτό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας. Ένα λεπτό διακοπή για να ξεπροβοδίσουμε τον Επίτροπο και θα συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα της ημερήσης διάταξης. Okay, okay. Thank you very much. Non me lo sopra. Ah? Okay, dear we uh, start. Ωραία. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, αρχίζουμε. Το επόμενο θέμα ανταλλαγή απόψεων με την ε, Ευρωπαϊκή ε, Υπηρεσία Ελέγχου και Δήλωση Νοσημάτων και έχει να κάνει με τον εμβολιασμό. Έχουμε διοργανώσει αυτή τη συνεδρίαση ε, ως εξής. Πρώτα μία παρουσίαση από τον προσκεκλημένο μας και αργότερα θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας δώσει τις δικές απόψεις και ακολουθεί η συζήτηση φυσικά. Αρχίζω αμέσως, θα δώσω το λόγο στον κύριο. Ποιος θα αρχίσει πρώτος. Κάτσε πολλό από ε, ε, ε, ε, η CDC να μας κάνει την παρουσίαση και μετά ο επόμενος ομιλητής. Ο κύριος Κάτσπολ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ όλους που μείνατε γιατί είναι πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό για τη δημόσια υγεία. Έχω τρία απλά μηνύματα να σας δώσω σήμερα. Τα εμβόλια έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα. Είναι πάρα πολύ ασφαλή και στην Ευρώπη δεν εμβολιάζουμε αρκετά τον πληθυσμό για να επιτύχουμε το επιθυμητό και το εφικτό αποτέλεσμα. Λοιπόν, στη σύγχρονη ιατρική και τα σύγχρονα εμβόλια ξεχνάμε πόσο ε, σημαντικές και σοβαρές είναι οι νόσοι που μπορούν να αποφευθούν με εμβόλια. Εδώ βλέπετε το Μαξ το 2004 ήταν ένα παιδί πάρα πολύ χαρούμενο και ε, ε, ε, δραστήριο και αθλητικό. Δυστυχώς uh, Δυστυχώς δεν τον εμβολίασαν και έπαθε η Λαρά που είναι μια σοβαρή ασθένεια και με επιπλοκές και το βλέπετε το 2012 και δυστυχώς λίγο μετά έχασε τη ζωή του ο Μαξ. Και αυτό μας θυμίζει ότι αυτές οι ασθένειες είναι πάρα πολύ σοβαρές και είναι και θανατηφόρες και προκαλούν πάρα πολύ σοβαρές ασθένειες ενώ μπορούν να προβληφθούν με εμβόλια. Και αυτό το μήνα είχαμε πάλι μια τέτοια υπενθύμηση με ένα πολύ ε, σοβαρό πρόβλημα διφθερίτιδας σε ένα εξάχρονο στην Ισπανία ανεμβολιαστό και ε, αυτό δεν μας θυμίζει απλώς πόσο σοβαρές μπορεί να είναι αυτές οι νόσοι, αλλά και πώς η απόκριση και η απάντηση είναι πάρα πολύ δύσκολη στη διαχείριση, ε, στη θεραπεία ε, για τη διφθερίτιδα, ας πούμε, χρειάζεται μια συγκεκριμένη αντιτοξίνη. Και ένα από τα γεγονότα που θα πρέπει να αναγνωρίσουμε είναι ότι αν δεν αλλάξει κάτι στο μέλλον, μπορούμε να ε, χάσουμε και τα αντιβιωτικά, δηλαδή να μην, να μην πιάνουν τα αντιβιωτικά, οπότε τα εμβόλια είναι όλο και πιο αποτελεσματικά για την πρόληψη. Όπως σας είπα λοιπόν οι εμβολιασμοί είναι πάρα πολύ αποτελεσματικοί και τα ίδια τα εμβόλια. Βλέπετε εδώ για την Ιλαρά την παροτίτιδα και την ερυθρά, με ποια ταχύτητα ε, μειώνεται ο αριθμός των κρουσμάτων από τη στιγμή που έχουν εισαχθεί τα εμβόλια. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση στη δημόσια υγεία που μέσα σε ένα με δύο χρόνια από την εισαγωγή των εμβολιασμών έχετε τέτοια τεράστια βελτίωση στη δημόσια υγεία. Και το θέμα δεν είναι ότι βλέπουμε λιγότερα κρούσματα παιδιών με ηλαρά, ε, ε, με παροτίτιδα, μαγουλάδες δηλαδή και ερυθρά δεν είναι μόνο αυτό, αλλά... Πω, πω, κοιτάξτε, η τεχνολογία δεν, δεν με Δεν ξέρω αν μπορείτε να τα διαβάσετε αυτά, αλλά βλέπουμε και πολύ λιγότερες περιπτώσεις σοβαρών, ε, Ισπανίων μεν, αλλά σοβαρών επιπλοκών. Ε, ε, σας είπα η εγκεφαλίτιδα από την Ιλαρά που έπαθε ο Μάξ ή ε, από την Ερυθρά, προβλήματα στην ακοή, παγκρεατίτιδα κτλ. Ε, υπάρχουν ε, λοιπόν πολύ αποτελεσματικές ε, μορφές παρέμβασης και αυτές είναι τα εμβόλια και είναι και επίσης και πάρα πολύ ασφαλή. Θα γνωρίζετε όλοι ότι με την πάροδο των ετών είχαμε κάποια προβλήματα, σκάνδαλα δημόσιας υγείας από το Ηνωμένο Βασίλειο που είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα με εμβόλιο τριπλούν ηλαράς παρατήτηδας ερυθράς και υποτίθεται ότι συνδέθηκε αυτό ε, με ε, αυτισμό. Αυτό έχει καταπέσει απολύτως ε, με επιστημονικά στοιχεία αποδεδειγμένα και στο τριπλούν έχει επανέλθει λοιπόν η εμπιστοσύνη, η λαράς παροτίτιδας ερυθράς και αρχίζει να εμβολιάζεται περισσότερο ο κόσμος και ο πληθυσμός. Τώρα έχουμε φάρμακα που είναι και πολύ ασφαλή και πολύ αποτελεσματικά. Παρόλα αυτά δεν καταφέρουμε να έχουμε τους στόχους ε, δημόσιας υγείας που είχαμε θέσει ε, και μπορούμε να φτάσουμε με τη χρήση αυτών των εμβολίων. Παράδειγμα, για την Ιλαρά είχαμε στόχους στην Ευρώπη ε, μέχρι το 2010 να εξαλειφθεί, το 2015 ακόμα έχουμε ούτε πρόκειται, το 2020 είναι ο ορίζον τώρα εξάλληψης και κρίση αυτής της νόσου. Και το πρόβλημα με την Ιλαρά είναι ότι τώρα έχουμε κρούσματα στη Γερμανία, στα γαλλογερμανικά σύνορα και σε άλλες χώρες, όπως βλέπετε εδώ, όπως σας δείχνω. Δυστυχώς ε, πέθανε ένα βρέφος στη Γερμανία από Ιλαρά και ε, μπορεί αυτό να επεκταθεί. Βλέπουμε κρούσματα και εξάρσεις στα σύνορα της Ευρώπης με πόλιο στη Συρία ε, είδαμε τεράστια κρούσματα ε, ηλαράς ε, και φυματίωσης στην Ουκρανία και σε άλλα μέρη του κόσμου. Υπάρχουν μεγάλες ταραχές και διαταράξεις των συστημάτων υγείας με νοσήματα που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Γιατί δεν έχουμε επιτύχει τους στόχους που είχαμε θέσει. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι η απροθυμία, αυτός ο δισταγμός να εμβολιάζονται. Και εδώ μπορεί να αφορά και τους επαγγελματίες υγείας και το κοινό. Κατά πόσο εμπιστεύονται το εμβόλιο, ότι είναι αποτελεσματικό, αυτό που γράφει πάνω, ας πούμε, αν ανταποκρίνεται, ή ζητήματα ασφαλείας, ε, αξιοπιστίας, ή μπορεί να είναι και θέματα Απλώς ότι δεν βολεύει κάποιος να πάει. Ας πούμε, ε, πρώτο κίνητρο είναι ο φόβος, σύμφωνα με κάποια έρευνα που κάναμε και μάλιστα ο βάσιμος φόβος και ο δισταγμός από τους επαγγελματίες υγείας, γιατί πολλές φορές δεν προσφέρουν αυτά τα εμβόλια, ενώ είναι φανταστικά και, και πάρα πολύ ασφαλή και προλαμβάνουν απόλυτα την ασθένεια. Βέβαια, ένα άλλος λόγος είναι ότι υπάρχουν πληθυσμοί που υποεξυπηρετούνται, που δεν έχουν πρόσβαση, που είναι μακριά για τις υπηρεσίες υγείας και δεν μπορούν να φτάσουν σε αυτές. Κοιτάξτε αυτές οι φωτογραφίες, βλέπουμε ορισμένες ομάδες, ε, παράτυπους μετανάστες Ρωμά και μετακινούμενες νομαδικές κοινότητες που πολλές φορές έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην πρόληψη, κοινωνικό αποκλεισμό γνωρίζουν, ένδια ή απλούστατα για λόγους ε, ε, ότι δεν είναι βολικό να φτάσουν. Έχουμε ένα πρόγραμμα δράσης ε, για την Ιλαρά και την Ερυθρά ε, με ιδιαίτερη εστίαση το ποια είναι τα στοιχεία και τι μπορεί να βοηθήσει για να φτάσουμε περισσότερο σε αυτούς τους πληθυσμούς. Τι γίνεται ας πούμε με τους αυτόχθονες πληθυσμούς που δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτούς. Αν ε, εντοπίσουμε τις αιτίε, ε, μπορεί αυτό να αφορά και τους μετανάστες και να επεκταθεί. Η Ευρώπη βεβαίω αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, όπως γνωρίζετε, όλο και περισσότερο. Τρίτον, υπάρχει ένα πρόβλημα προμήθειας εμβολίων. Σήμερα στην Ευρώπη έχουμε πραγματικές δυσκολίες να βρούμε εμβόλια ιδιαίτερα το εμβόλιο για την προστασία ε, κατά του κοκκίτη. Το 1 τρίτο των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δηλώσει δυσκολία να βρουν εμβόλιο κοκκίτη. Γιατί ε, ε, εδώ υπάρχει ένα συνδυασμό παραγόντων. Υπήρχε πρόβλημα στη διαδικασία παραγωγή από ορισμένου παρασκευαστέ και έχει αυξηθεί και η ζήτηση. Γιατί πολλέ χώρε έχουν νέα προγράμματα εμβολιασμού εγγύων για να προστατεύονται τα νεογέννητα τους πρώτους μήνες ζωής. Δηλαδή υπάρχει και αυξημένη ζήτηση και πρόβλημα στην παραγωγή, οπότε υπάρξει ένα θέμα έλλειψης ε, εμβολίων κοκκίτη. Επίσης, τρία από, τρεις από τους εννιά μεγάλους ε, παραγωγείς εμβολίων αντιγρυπικών έκλεισαν. Σταμάτησαν να παράγουν. Λοιπόν, τι κάνουμε εμείς στο κέντρο δήλωσης και ελέγχου νοσημάτων. Ε, έχουμε μια διαπιστημονική προσέγγιση και φέτος στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε ε, ε, ε, με βάση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ανοσοποίηση, να φτάσουμε σε ομάδες που διστάζουν, να ανταλλάξουμε ε, γνώσεις και απόψεις για να ενισχυθούν ε, τα προγράμματα εμβολιασμού. Είναι το έργο Βένης, Βενετίας, ένα δίκτυο για νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό και αν χρειαστεί και επιτόπιες επισκέψεις στα κράτη-μέλη για να δίνουμε συμβουλές και οδηγίες. Γενικά λοιπόν θέλουμε να υποστηρίξουμε την πρόληψη τον έλεγχο των νοσημάτων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Ε, σας λέω προλαμβάνουμε, προκαταλαμβάνουμε κάποια συμπεράσματα του Συμβουλίου, αλλά από το 2011 υπάρχουν συμπεράσματα του Συμβουλίου που είναι εξίσου επίκαιρα σήμερα, κάθε λέξη τους. Και θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα που σας είπα, το, δισταγμό του κόσμου, ε, πληθυσμούς που δεν έχουν πρόσβαση και ε, χάσματα και κενά στην ανοσοποίηση και στην ανοσία του πληθυσμού. Ε, και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε μια σειρά κατευθυντηρίων γραμμών και οδηγιών και θα πρέπει να είναι αξιόπιστα και ισχυρά τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και για την προσοχή σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα πάμε στον επόμενο μιλητή. Πάμε στο Μπόι Κύριε Μπερτολίνη, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Λαβία. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μιλήσουμε για τους εμβολιασμού. Πρόκειται για έναν από τους πιο σημαντικούς τρόπους παρέμβασης που έχουμε στη δημόσια υγεία. Τι θα κάνω σήμερα, εν συντομία. Θα σας συνοψίσω κάποια από τα ζητήματα τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί και από το συνάδελφο και θα επεκταθώ λίγο στον τομέα των παρεμβάσεων και των δράσεων που προτείνει η ΠΟΗ σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ανοσοποίησης ε, ε, στις χώρες του ΠΟΗ και φυσικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε ότι ο εμβολιασμό είναι ε, ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για τη δημόσια υγεία και γνωρίζουμε επίση ότι αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο η ανθρωπότητα κατάφερε να εξαλείψει πριν από κάποιε δεκαετίε ε, από προσώπου γης ε, μία από τις πιο θανατηφόρες ασθένειες οι οποίες επηρέασαν ε, τις ε, προηγούμενες γενιές, την ευλογιά. Και πλησιάζει επίσης και στην εξαφάνιση της πολιομιαλίτιδας. Και θα ήθελα εδώ επί τη ευκαιρία να ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει τις προσπάθειες που κάνουμε σε κάποιες χώρες, τις σύστατες προσπάθειες για να εξα... εκριζώσουμε και αυτή την ασθένεια που είναι πάρα πολύ σοβαρή. Υπάρχουν όμως αρκετά πράγματα ε, τα οποία πρέπει να σκεφτούμε όσον αφορά στο ερώτημα γιατί θα πρέπει να εμβολιάσουμε. Πρέπει ε, καταρχάς να σκεφτούμε ότι είναι δικαίωμα των ανθρώπων να προστατεύονται από αυτές τις ασθένειες. Είναι ένας πολύ αποτελεσματικός μηχανισμός και αν δείτε τα αριθμητικά στοιχεία εκτιμούμε ότι 13,8 ε, εκατομμύρια θάνατοι έχουν προληφθεί στον τομέα, ε, στην, συγγνώμη, στην περιοχή της Ευρώπης του, της ΠΟΗ της Ρωσίας που σημαίνει ότι ε, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Επίσης υπάρχει και η σχέση κόστους αποτελεσματικότητας. Βλέπετε εδώ στη διαφάνεια έχουμε στοιχεία από μια πρόσφατη μελέτη για τον εμβολιασμό για το HPV, το παπιλώμα βούρους, ένα πρόσφατο εμβόλιο εκτιμάται ότι ε, εάν εμβολιαστούν 58 εκατομμύρια 12χρονα κορίτσια σε 179 χώρες θα υπάρξει πρόληψη 690.000 περιπτώσεων ε, ε, καρκίνου της μήτρας και 420.000 ε, θάνατοι, του τραχύλου συγγνώμη, της μήτρας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική πληροφορία σε ένα κόστος το οποίο εκτιμάται στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια αλλά αν δούμε την ανάλυση κόστους αποτελεσματικότητας είναι πάρα πολύ επωφελές δεδομένου ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλά για να θεραπευτούν οι γυναίκες οι οποίες πάσχουν από τη συγκεκριμένη νόσο έχουμε και κάποια στοιχεία όσον αφορά την κάλυψη για τον εμβολιασμό στην Ευρώπη. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε ε, ένα καταμερισμό αναχώρα. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποιες εξ αυτών. Υπάρχουν αρκετές διαφορές στην Ευρώπη ε, σε σχέση με το ε, στόχο του 95% του εμβολιασμού για την Ιλαρά. Στην Γαλλία έχουμε 67% κάλυψη, στην Αυστρία 64% και έχουμε χώρες οι οποίες Απ' την άλλη πλευρά ε, είναι πολύ κοντά στο 95, κάποιες το έχουν πετύχει, για παράδειγμα η Σουηδία ή και άλλες χώρες. Το σημερινό λοιπόν κενό το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουμε είναι κενό το οποίο θα πρέπει να το συμπληρώσουμε ε, ενώπιον και στεναρών αντιστάσεων από κάποιες ομάδες, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αποδείξεις που καταδεικνύουν αυτό το οποίο πολύ σωστά παρουσίασε ο συνάδελφος προηγουμένως. Υπάρχει ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Ε, έχετε εδώ αυτό το οποίο ανέφερε και ο συνάδελφος προηγουμένως, οι συνέπειε της μελέτης η οποία ανακλήθηκε. για τη σχέση μεταξύ αυτισμού και ηλαράς, που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Και εδώ βλέπετε όταν δημοσιεύθηκε η μελέτη ε, ότι μερικά χρόνια αργότερα η κάλυψη της, ε, του εμβολιασμού στην Ιλαρά στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε μια πτώση και χρειάστηκαν χρόνια για να ξανανεύει στα προηγούμενα επίπεδα. Αυτή είναι λοιπόν πάρα πολύ σοβαρή συνέπεια. Θα πρέπει να μπορούμε να την κατεμπαλοποιήσουμε με αποδείξεις, ε, με πάθος και με δράση φυσικά. Και αυτό είναι αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα. Εδώ έχουμε την καμπύλη του εμβολιασμού για τη γρήπη στην Ιταλία. Ο στόχος για τα άτομα 65 ετών είναι περίπου 75% και βλέπετε ότι από το 2009-2010 ε, ε, η κάλυψη σε σχέση με το στόχο πήγε από το 65% στο 49%. Και πέρσι, την τελευταία εποχή δηλαδή, ε, είχαμε και άλλη μείωση λόγω μιας λανθασμένης φήμης ότι το εμβόλιο κατά της γρήπης ε, σχετίζεται με θανάτους ηλικιωμένων ατόμων, κάτι το οποίο δεν αποδείχθηκε. Επομένως αυτές οι φήμες επηρεάζουν και νέους αλλά και ηλικιωμένους. Εδώ στο διάγραμμα συνοψίζουμε κάποια από τα στοιχεία τα οποία είχαμε τα τελευταία χρόνια, διάφορα κρούσματα και επιδημίες οι οποίες υπήρξαν για αρκετούς λόγους που αναφέρθηκαν ήδη και καταδεικνύουν ότι ένα από τα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε με ασθένειες τις οποίες μπορούν να προλάβουν τα εμβόλια είναι ότι δεν είναι ε, διαβίου αυτή η πρόληψη. Πρέπει να υπάρξουν και άλλες δράσεις και αυτές οι δράσεις για τον εμβολιασμό μπορεί να μην έχουν καμία αξία από πλευράς επικοινωνίας. Δεν είναι είδηση. Όταν ένα εμβόλιο είναι αποτελεσματικό δεν υπάρχουν επιχαίοι τίτλοι σε εφημερίδες γιατί κανείς δεν έχει πρόβλημα. Και αυτό φυσικά δημιουργεί πρόβλημα διότι μειώνεται η προσοχή της ε, ε ποιότητας ε, των όσων χαράζουν πολιτική, των ηθινόντων και του ε, κοινού φυσικά. Πρέπει να υπάρχει συνεχής ενημέρωση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο συνάδελφος αναφέρθηκε για παράδειγμα σε κάποια κρούσματα ηλαράς, αλλά ε, το 2007 είχαμε 7.000 περιστατικά ηλαράς και ε, διπλασιάστηκαν το 2014. Και αυτό αναφέρεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όταν έχουμε κρούσματα. Όταν όμως δεν έχουμε κρούσματα τότε δεν υπάρχει πρόβλημα και επομένως μειώνεται και η προσοχή του κοινού και υπάρχουν και άλλες πτυχές οι οποίες δεν ε, ε, ε τις φροντίζουμε καταλήλως ακριβώς γι' αυτό. Ήδη είπαμε ότι ο στόχος της εκρίζωσης της ηλαράς ε, στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια μέχρι το 2020 είναι πλέον μεταξύ ε, του προγράμμα, των στόχων του προγράμματος δράσης για τον εμβολιασμό. Θα σας πω δύο λόγια παραπάνω στη συνέχεια και εδώ σε κόκκινο έχουμε τις περιοχές τις οποίες ακόμα ευδοκιμεί η λαρά και βλέπουμε ότι ε, είναι ενθυμική σε κεντρικά ε, περιοχές της Τουρκίας, της Ρωσίας. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αρκετές χώρες. Η ΠΟΗ συστήνει ένα κατάλογο εμβολίων. Εδώ έχουμε τον κατάλογο των εμβολίων που προτείνουμε. δεν υπάρχουν όλα αυτά τα εμβόλια στις διάφορες χώρες της Ευρώπης. Εδώ βλέπετε ποιες ε, χώρες έχουν, ε, ε, βάλει, έχουν εισαγάγει εμβόλιο για τον πνευμονόκοκο. Εδώ έχουμε το HPV. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Όταν η κάλυψη εμβολιασμού για κάποιες περιπτώσεις διαφέρει σε διάφορες χώρες, η κυκλοφορία του ιού είναι πολύ υψηλή και αυτό μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα σε χώρες στις οποίες υπάρχει μεν εμβολιασμός αλλά δεν χρησιμοποιείται ευρέως. Τώρα, πολύ σύντομα, για να μην καθυστερήσουμε, σίγουρα υπάρχει έκκληση για να υπάρξει μεγαλύτερη δέσμευση για νοσοποίηση και φυσικά θα πρέπει να εγκριθεί και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τον Εμβολιασμό το, 2012, το 2014, συγγνώμη, το οποίο πρόγραμμα έχει ένα όραμα. Το όραμα είναι να υπάρχει ε, μια ζώνη τρία για ε, νόσους οι οποίες μπορεί να προληφθούν από τον εμβολιασμό, δηλαδή να υπάρχουν ασφαλή ε, ε, εμβόλια σε προσιτές τιμές διαθέσιμα για όλους και εδώ δεν θα ήθελα να επισέλθω σε λεπτομέρειες και να σας κουράσω, αλλά αυτό διαρθρώνεται σε έξι βασικούς στόχους, για παράδειγμα να ε, παραμείνει ε, η κατάσταση ε, στην οποία δεν υπάρχει πολεμιολίτιδα και να εξαφανιστεί η Λαρά και η Ερυθρά. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δεσμευτούν όλες οι χώρες να είναι προτεραιότητα εμβολιασμό στις συγκεκριμένε δράσεις. Αυτό είναι ο στόχος 1 για παράδειγμα και ο στόχος 2 είναι να κατανοήσουν οι άνθρωποι την αξία της ανοσοποίησης και των εμβολίων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξουν μια σειρά από δράσεις για να επιτευχθεί ο στόχος. Τέλος, το πρόγραμμα δράσης το οποίο εγκρίθηκε από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Επικράτης, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γνωρίζετε, οι δεσμεύσεις της ΠΟΗ δεν είναι δεσμευτικές, είναι με πολιτικές δεσμεύσεις, ε, αλλά ε, ε, δεν είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και εδώ έχουμε κάποια από τα στοιχεία τα οποία ε, δεν μας επιτρέπουν να έχουμε αποτελεσματική εφαρμογή του εμβολιασμού. Καταρχάς δεν υπάρχει ε, δέσμευση σε κάποιες χώρες. Επομένως θα πρέπει να διασφαλίσουμε να υπάρχει δέσμευση. Υπάρχουν κάποια κενά ανοσίας, αυτό το αναφέραμε, η κάλυψη που πρέπει να υπάρξει, ο στόχος που, πρέπει, που έχει καθοριστεί από κάθε χώρα και από την ΠΟΗ. Επίσης, το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις για τα εμβόλια και κάποιοι δεν θέλουν να εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Πρέπει να υπάρξει κατάλληλη εκστρατεία ενημέρωσης και υποστήριξη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να μας υποστηρίξουν και πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις. Και πάλι ε, επαναλαμβάνω ότι όταν είναι αποτελεσματικά τα εμβέλια, δεν αποτελούν είδηση. Επομένως ε, ε, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι πρώτες λανθασμένες πληροφορίες που μπορεί να κυκλοφορήσουν για να αλλάξουμε άποψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στον εμβολιασμό ο εμβολιασμός μάλλον να ε, ενταχθεί στα συστήματα υγείας και να είναι από τα ε, τσεκά που γίνονται και επίσης είναι πολύ σημαντικός ο εμβολιασμός και για τους μετανάστες γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη μείωση της κυκλοφορίας των ιών και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν κατάλληλες πληροφορίες και να αναφέρονται όλα τα περιστατικά. Ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ α ρωτήσουμε όμω τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Άνταμ, που είναι ε, αναπληρωτή μετάρχη στην ε, Μονάδα Υγείας ε, της αρμόδια Γενικής διεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα καταρχήν να τονίσω ότι ο Επίτροπος Ανδριοκάητες αποδίδει ύψιστη προτεραιότητα στο θέμα του εμβολιασμού. Είναι για τον Αρμόδιο Επίτροπο πολύ σημαντικό θέμα και όπως αναφέρθηκε από τους προλαλήσαντες, με τον εμβολιασμό έχουμε πολύ ισχυρό εργαλείο και μάλιστα πιάνουν τόπο και τα χρήματα. Έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα από άποψη ε, κόστος ωφέλους. Όλοι τα στοιχεία έδειξε το τεράστιο δυναμικό των κατάλληλων προγραμμάτων εμβολιασμού. Αυτό που διαπιστώνουμε όμως και αναφέρθηκε και όλα είναι ότι έχουμε και κάποιες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Μία από αυτές αφορά το γεγονός ότι η ε, πολιτικοί θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων εμβολιασμού και στην <clears throat> αξιολόγηση της αποτελεσματικότητά τους. Ε, επίσης θα πρέπει να εξηγήσουμε καλύτερα ε, και να επικοινωνήσουμε καλύτερα σχέση με τα πλεονεκτήματα του εμβολιασμού. Βέβαια το θέμα του εμβολιασμού είναι εθνική αρμοδιότητα. Αυτό που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να στηρίξει τα κράτη-μέλη και αυτό το κάνουμε οργανώνοντας εκδηλώσεις για την αύξηση της ε, ευαισθητοποίησης, ε, την ανταλλαγή των πληροφοριών. Χρηματοδοτούμε μελέτες ε, σχετικές και ενημερώνουμε για την κατάσταση των πραγμάτων και της εξέλιξης. Και φυσικά το έργο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Όσων μας ε, στηρίζει με την εμπειρογνωμοσία, με την ε, επαγρύπνηση και την καθοδήγηση προς τα κράτη-μέλη. Κάτι άλλο που κάνουμε είναι συζητούμε με τα κράτη-μέλη στην ε, Επιτροπή Ασφάλειας της Υγείας με βάση το άρθρο με τον κανονισμό 182. συζητούμε λοιπόν σε αυτή την Επιτροπή όταν η ΠΟΗ θεώρησε την πολιομελίτιδα ως διεθνή ε, ε, επίγουσα ανάγκη αντιμετώπισης, προσπαθούμε να συντονίσουμε τις δραστηριότητες και τα μέτρα μας. Και αυτό που συζητούμε με τα κράτη-μέλη, αυτό που συζητήσαμε τον Απρίλιο, ε, είναι τι γίνεται με την έλλειψη που διαπιστώνουμε στα, στην προμήθεια εμβολίων, για παράδειγμα το εμβολίο κοκκίτι όπως μας είπε ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων. Ε, μας ενδιαφέρουν και πληροφορίες ε, για την κατάσταση της εφαρμογής ό,τι αφορά τις συστάσεις ε, του Συμβουλίου. Για παράδειγμα, για τη γρήπη την εποχιακή, προσπαθήσαμε ε, να δούμε τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Διαπιστώσαμε ότι δεν υλοποίησαν όλοι τα κράτη-μέλη τους στόχους. Υπάρχει χαμηλή κάλυψη με το αντιγρυπικό εμβόλιο. Και επίσης σκεγγραφούμε τα μελλοντικά βήματα και υποβάλλουμε προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης. Γι' αυτό και τον Απρίλιο οργανώσαμε μια διάσκεψη με συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων προκειμένου να συζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι με τα κράτη-μέλη τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η κάλυψη με εμβόλια. Και συμπέρασμα του σημενερίου είναι ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν προς το στόχο αυτό, να βελτιώσουν την κάλυψη του εμβολιασμού, να θεσπίσουν εθνικά πλαίσια, να καθορίσουν κανόνες και ευθύνες και επίσης να εξασφαλίσουν ε, την πολιτική, την εφαρμογή των προγραμμάτων προγραμματισμού, να παράσχουν ε, εμβολιασμό, να παρακολουθήσουν την λήψη και αποτελεσματικότητα των εμβολίων και να προβούν και σε αναθεώρηση σε περίπτωση που διαπιστώνονται κενά ή θεωρούνται κάποιες δράσεις ως ακατάλληλες. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι να ενισχύσουμε τις δραστηριότητες κοινοποίησης και ενημέρωσης και προς τους ε, νομοθέτες και προς τους ε, επαγγελματίες ε, στον τομέα της υγείας. Αλλά θα πρέπει να ενημερώνουμε και το ευρύ κοινό για τα ωφέλη του εμβολιασμού. Δεδομένων όλων αυτών των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, Χαιρετίζουμε ιδιαίτερως ε, ε, την υιοθέτηση από το Συμβούλιο το Δεκέμβριο των συμπερασμάτων του γιατί έτσι φέρνουμε το θέμα του εμβολιασμού στο επίκεντρο της προσοχής. Οι στάση του Συμβουλίου ζητούν στενότερη συνεργασία και βελτίωση των εθνικών προγραμμάτων εμβολιασμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κρατημέλη καλούνται να συνεργαστούν για να αναπτύσσουν κοινά προγράμματα δράσης, να αξιοποιήσουν τις βέλτιστες πρακτικές και να βελτιώσουν την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων εμβολιασμού. Γιατί όπως είπε ο κ. Κάτσπολ υπάρχουν κενά και στην ε, εποπτεία και στο feedback. Δεν γνωρίζουμε πώς εφαρμόζεται σε πολλές περιοχές ο εμβολιασμός και κατά πώς εφαρμόζεται. Οπότε με βάση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου φροντίζουμε να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για να στηρίξουμε τα κρατη και φυσικά στενιζόμαστε τους ε, στόχους της ΠΟΕ στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τον Εμβολιασμό. Και επιπλέον προσπαθούμε να θαρρύνουμε τα κράτη-μέλη στις προσπάθειές τους να ανταλλάσσουν πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και βέλτιστες πρακτικές και να τα εψυχώσουμε να εστιάσουν και στην παρακολούθηση ε, των προγραμμάτων. Αυτά και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε ώρα για συζήτηση. Θέλει κάποιο ευρωβουλευτή ε, το λόγο να υποβάλει ερωτήσει. Κυρία Κάντεμπαχ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι λιγότερο ερώτηση. Θα ήθελα πραγματικά να σα ευχαριστήσω γιατί τα τελευταία χρόνια και σε σχέση με τους εμβολιασμού και ε, για τα παιδιά έχουμε κάνει πολλές κοινέ ε, ε, διοργανώσεις με την ΠΟΗ, την ECDC και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πραγματικά πρέπει να πω ότι έχουν γίνει ε, τεράστιες προσπάθειες και πάρα πολύ εντατικές. Και ξέρετε ότι πολλές φορές πέφτει κανείς θύμα της επιτυχίας του. Υπάρχει μια κόπωση ανεξήγητη των εμβολιασμών και αυτό είναι ε, θύμα της επιτυχίας. Όπως είπατε, όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά ούτε είδηση είναι ούτε φαίνεται. Ε, όταν κάτι πάει στραβά τότε είναι είδηση. Και το γεγονός ε, ότι πρέπει να κάνουμε προσπάθειες και είμαστε στο σωστό δρόμο είναι καλό. Εσείς τι θέλετε από εμάς τους Ευρωβουλευτές για να υποστηρίξουμε τις δικές σας προσπάθειες. Τι μπορούμε να κάνουμε για σας. Ε, έχουμε ένα κοινό στόχο. Ο εργαλειασμός είναι ένα εργαλείο το οποίο όχι απλώς σώζει ζωές, αλλά και σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας. Πρέπει να αποδείξουμε ότι για κάθε εμβολιασμό ε, υπάρχει λόγος. Θα πρέπει να το στοιχειοθετούμε με αριθμούς και στοιχεία για να μην μπορεί κανείς να επικαλεστεί την οικονομική κρίση το πρόβλημα. Δυστυχώς στην πολιτική σήμερα καταλαβαίνουν περισσότερο από αριθμούς και λιγότερο από τα γενικά που λέμε για τη δημόσια υγεία. Θα σας παρακαλούσα να μας δώσετε περισσότερο υλικό για να μπορέσουμε να στοιχειοθετήσουμε και εμείς τις απόψεις μας, για να βοηθήσουμε και τους υπόλοιπους εμβολιασμούς. Thank you very much, uh, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριο Σεκχάουτ. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ για αυτό το μακροσκελές διαφημιστικό υπέρ του εμβολιασμού. ξέρουμε και ποιοι είναι οι σπόνσορες, οι χορηγοί. παροτρύνεται για ενίσχυση του εμβολιασμού. Αλλά πολλές επικρίσεις ακούγονται και πολλές ανησυχίες ε, προβληματίζουν το κοινό και αυτές θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη. Έχω την αίσθηση ότι τέτοιες εκκλήσεις ε, ε, για να διορθωθεί με εκστρατείες αυτή τη διστακτικότητα για το εμβόλιο είναι σαν να μην λαμβάνεται σοβαρά υπόψη αυτά τα, αυτές τις ανησυχίες του κοινού. Βέβαια, ήταν σαφέστατο το παράδειγμα, αλλά υπάρχουν και άλλες ανησυχίες. Πώς θα τις αντιμετωπίσετε. Για παράδειγμα, Υπάρχει ένα εμβολιασμό για το, για το, καρδεζ, το, το εμβόλιο Καρδεζίλ. Τι θα κάνετε ε, προκειμένου να αναπτυχθούν εναλλακτικέ λύσεις. Ε, όχι μόνο να ε, οθείτε για πράγματα κατηγορώντας το κοινό ότι κάνει λάθος ή το διαδίκτυο ότι κάνει λάθος. Πώς θα βρούμε ασφαλείς εναλλακτικέ λύσεις. Για παράδειγμα για το εμβόλιο Γκαρντασίλ αναφέρθηκε ότι περιέχει αλουμίνιο. Φυσικά δεν θέλει να παίρνει κάτι τέτοιο ο κόσμος. Γιατί δεν βρίσκεται εναλλακτικέ, γιατί δεν μεριμνάτε και για αυτά τα θέματα. Κάτι που με ενοχλεί είναι ότι κανένας ομιλητής δεν μα είπε για την κατάσταση στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Εκεί διαπιστώνουμε ότι τα λοιμώδη νοσήματα αυξάνονται αυτή τη στιγμή. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει και να ανησυχεί ε, θεσμούς όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Τι θα κάνουμε γι' αυτό, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στην Ελλάδα για να μην επιδεινωθεί η κατάσταση. Μόνο για εμβόλια μας είπατε να τα προωθήσουμε, ε, να τονώσουμε την χρήση τους, αλλά ε, όργανα όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων θα πρέπει να αναλαμβάνει υπόψη και άλλα θέματα, τα προβλήματα στην Ελλάδα και να επισημαίνει ότι αυτά θα πρέπει να διορθωθούν. Όχι να επικεντρώνεται στα εμβόλια που χρειαζόμαστε, αλλά και σε άλλες πολιτικές. Κύριος Ντεμέσμακερ, δύο σύντομες ερωτήσεις, μικρές ερωτησούλες. Είπατε ότι υπάρχει πρόβλημα με την παραγωγή ορισμένων εμβολίων τι σπταίει, είναι οικονομικά τα προβλήματα, πρακτικά, τι είδους είναι. Και μια δεύτερη μικρή παρατήρηση ερωτησούλα, μιλήσατε για την έξαρση ορισμένων ε, ε, λιμωδών ε, ή μεταδοτικών ασθενειών στα εξωτερικά μας σύνορα. Αναφερθήκατε μάλιστα και στην Ουκρανία. Ανησυχώ πάρα πολύ, έχω θορυβηθεί, γιατί έχω πάει πολλές φορές στην Ουκρανία Μιλάτε για πολιομιελίτιδα, για ηλαρά και όλες, ακόμα και για φυματίωση. Μα τι έγινε, έχει καταρρεύσει ήδη ή καταραίει το σύστημα υγείας στη χώρα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, πρώτα για τους ίδιους τους Ουκρανούς, αλλά και για μας. Ε, γνωρίζοντας ότι είναι λιγότερο από τρει ώρες η πτήση Βρυξέλλες-Κίεβο. Και εμείς τι θα κάνουμε λοιπόν γι' αυτό. Thank you, ε, κύριε Γκρότε, ευχαριστώ πολύ. Καταλάβαμε λοιπόν για ποιο λόγο κάνουμε αυτή την οργάνωση, γιατί υπάρχει ένα κενό και τρύπες στο δίκτυο ε, εμβολιασμού ε, και στη χώρα μου υπάρχει μια κόπωση εμβολιασμών και οι διάφορες θεωρίες συνωμοσία οργιάζουν ότι καλύτερα να μην εμβολιάζει τα παιδιά σου, μην πάθουν και τίποτα. Και πολύ ωραία μας είπατε ε, τι ε, έχει γίνει με μεμονωμένους ασθενείς. Εμένα τι με ενδιαφέρει να ρωτήσω. Το 2013 είχαμε μια οδηγία για επικίνδυνα διασυνοριακά κρούσματα. Ε, είναι μια οδηγία που λέγεται 2013 18. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι κάνει ε, και πώς συνεργάζεται με το ECDC και με τον ΕΟΦ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Υπάρχει συνεργασία, συντονισμός για να προχωρούν καλύτερα τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον εμβολιασμό, βεβαίως ο καθένας μπορεί να ανοίξει τα σχέρες του και να πει είναι θέμα των κρατών μελών. Υπάρχει όμως καμιά δυνατότητα από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αλλά και από τον Οργανισμό για τον έλεγχο και την πρόληψη των νοσημάτων να προχωρήσουμε και ανέπως. Ναι, και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για να το εξασφαλίσουμε αυτό. Έτσι ώστε το ποσοστό των εμβολιαζομένων να αυξηθεί και να αυξηθεί και η ανοσία για όλους. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί εδώ διαπληκτιζόμαστε και, και ε, όλες οι πολιτικές ομάδες μάλλον διαρριγνύουν τα μάτια τους ότι πρέπει να μειώσουμε τη χρήση αντιβιωτικών και εκεί που θα μπορούσε να γίνει αυτό πολύ απλά με εμβολιασμό και ανοσία ε, δυσκολευόμαστε και προβληματιζόμαστε. Σας ευχαριστώ και πάλι για αυτό που είπατε και για την παρουσίαση, κύριε Κάθχο. Thank you very much, Mr. Pedicini. Pedicini. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω τρεις ερωτήσεις και ελπίζω να είμαι σύντομος. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε εδώ για να ε, κάνουμε συνδικαλισμό για τη χρησιμότητα των εμβολίων. Γνωρίζουμε ότι κάποια ήταν ιστορική σημασία και πραγματικά έσωσαν ανθρώπινα ζωέ ε, ε, διότι έσωσαν από κάποιες ασθένειες όπως η πολιομελίτιδα, ο τέτανο, η απατήτιδα β και η διφθυρίτιδα. Εκείνο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί κάποια εμβόλια είναι υποχρεωτικά σε κάποιες χώρες και προαιρετικά σε κάποια όλα. Ε, διότι ε, είναι γνωστά τα εμβόλια και ανανόσο σε κάθε χώρα. Είναι δυνατόν να διευκρινίσουμε τη σχέση μεταξύ κρουσμάτων και κάλυψης εμβολιασμών, ειδικώ ε, για χώρες που γνωρίζουμε ότι δεν προβλέπεται υποχρεωτικός εμβολιασμός και τι αποτελέσματα έχουμε για τις χώρες που είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός. Δεύτερη ερώτηση. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται στις χώρες στις οποίες ε, δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, αλλά για το παράδειγμα της Ιταλίας. Στην Ιταλία έχουμε τέσσερα υποχρεωτικά εμβόλια στα μικρά παιδιά, αλλά ε, δίνεται τυπικά και ένα εμβόλιο το οποίο περιλαμβάνει και δύο προαιρετικά ε, εμβόλια για το κοκκίτι και για την γρήπη τύπου Β. Ε, δεν διατίθενται όμως αυτά τα εμβόλια μεμονωμένα και αυτό κατά την άποψή μας είναι πολύ σημαντικό διότι αυτή η πολλαπλή χορήγηση των εμβολίων μπορεί να δημιουργήσει και σοκ στο νοσοποιητικό σύστημα. Επομένως, από οικονομική σκοπιά καταρχάς η διαδικασία ε, έχει μια μεγαλύτερη δαπάνη η οποία είναι περιττή και με την οποία επιβαρύνεται το κράτος και έχουμε παραπάνω 115 εκατομμύρια το χρόνο δαπάνη για αυτό το σκοπό υπάρχουν μέτρα σε κάποιες χώρες που θα μπορούσαμε να περιορίσουμε ε, αυτή την κατασπατάληση των δημοσίων κονδυλίων και επίσης ε, μήπως είναι πολύ μεγάλος ο κατάλογος των εμβολίων. Πολλές φορές ε, μας λέγεται ότι πρόκειται για παρεπίπτουσες ζημίες που εμφανίζονται σε πολύ μικρά ποσοστά όπως γίνεται και με παρενέργειες που έχουμε για φάρμακα κοινή χρήσης. Ορισμένες φορές υποχρεούνται όμως όλος ο πληθυσμός να λάβει κάποια εμβόλια. Σε ποιο βαθμό λοιπόν οι γονείς είναι κατάλληλοι ενημερωμένοι για τις παρενέργειες που μπορεί να υπάρξουν από τα εμβόλια και πώς μπορούμε ε, να δείξουμε ποιες είναι οι ε, πραγματικές ε, επιστημονικές ενδείξεις για τα εμβόλια όταν οι ίδιες οι φαρμακευτικές εταιρείες δίνουν χρήματα για τις έρευνες αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε πολλές ερωτήσεις και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις απαντήσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και για τις ερωτήσεις σας. Προσπάθησα να τις καταγράψω. Ευχαριστώ για την ερώτηση το πώς μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βοηθήσει. Σίγουρα η προβολή της ε, αξίας που έχουν τα εμβόλια, εμβολιασμοί για τη δημόσια υγεία είναι πολύ σημαντικό. Επίσης παρακολούθηση των εμβολιασμών. Εκεί θα μπορούσατε να συνδράμετε με πιο συγκεκριμένο τρόπο ή να εξετάσετε τρόπους ε, με τους οποίους ε, θα αναλάβετε πρωτοβουλίες για να φτάσουμε σε πληθυσμούς και ομάδες πληθυσμών που υποεξυπηρετούνται. Εκεί θα είναι σημαντική η αξία και η συμβολή σας. Σε ό,τι αφορά την απάντηση ε, του προτελευταίου συναδέλφου, το άνοιγμα και η διαφάνεια είναι πολύ σημαντικά θέματα πολύ ευχαριστώ ε, να επανέλθω ε, για να συζητήσουμε, να αφιερώσουμε ολόκληρη συνεδρίαση για το τι κάνουμε στην Ελλάδα και αλλού. Αλλά το θέμα το σημερινό ήταν τα εμβόλια, οι εμβολιασμοί. Γι' αυτό μίλησα για τους εμβολιασμού. Πολύ ευχαρίστω να έρθω άλλη στιγμή και να σας μιλήσω για τη σημασία που δίνουμε στην Ελλάδα ε, και σε άλλες χώρες και πώς βοηθούμε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Το άνοιγμα και η διαφάνεια φυσικά που θα στηρίζονται σε ε, τεκμηριωμένα επιστημονικά πορίσματα, γιατί υπάρχει καλή και κακή επιστήμη. Είχαμε μία ανακριβή μελέτη. Αυτό είναι κακή επιστήμη. Θα πρέπει να προβάλλουμε τα σωστά επιστημονικά πορίσματα. Για το αλουμίνιο και το σχετικό εμβόλιο. Το αλουμίνιο χρησιμοποιείται σε εμβόλιο από τότε που ξεκίνησαν τα εμβόλια. Δεν υπάρχει μία απόδειξη ότι είναι επιβλαβές. Είναι σημαντικό συστατικό του εμβολίου ε, το αλουμίνιο, γιατί βελτιώνει την ε, αποτελεσματικότητά του. Χρειαζόμαστε όμως ε, ανοιχτά, αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τη χρήση του αλουμινίου. Τώρα, γιατί υπάρχουν τα προβλήματα με το κοκκίτι και με το σχετικό εμβόλιο. Υπήρξαν πρακτικά προβλήματα παραγωγής από ό,τι ξέρω Πρακτική φύση ήταν τα προβλήματα για το ότι σταμάτησε το εμβόλιο κοκκίτη, η παραγωγή του. Και τέθηκε και μία ερώτηση για το πώς μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο σε, τους, σε αυτές τις ομάδες που υποεξυπηρετούνται. Καταρχήν θα πρέπει να φροντίσουμε όταν έχουμε καλές αποδείξεις για το τι λειτουργεί να το, και το γνωρίζουμε να το προβάλλουμε να γίνεται σωστή επικοινωνιακή χρήση. Στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, είχαμε πρωτοπόρο καταπληκτικό έργο για διαμεσολαβητές που μεσολάβησαν στην κοινότητα Ρωμά και υπήρχε σημαντική πρόοδος. Ελπίζω το παράδειγμα της Βουλγαρίας να το ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Μπορούμε να συγκρίνουμε την κάλυψη των εμβολιασμών με τη συχνότητα των κρουσμάτων. Ναι. Και επίσης έχουμε πολύ ξεζητημένα μαθηματικά μοντέλα που δείχνουν ποιο, τι επίπεδο ε, κάλυψης εμβολιασμού μπορεί να εμποδίσει τη μετάδοση. Υπάρχει και σχετική επιστημονική βιβλιογραφία εκτεταμένη. Ε, μίλησαμε για το αντιγρυπικό εμβόλιο, για το εμβόλιο της ιλαράς και το στόχο κάλυψης ε, με εμβολιασμό για την ΙΛΑΡΑ. Και αυτά τα στοιχεία στηρίζονται σε τεκμηριωμένες και άρτιες μελέτες που ε, λένε τι ε, επίπεδο κάλυψη χρειάζεται για να εμποδιστεί η μετάδοση. Τώρα, πώς θα επιτύχουμε αυτά τα επίπεδα, αυτό είναι άλλη συζήτηση, άλλο Ευαγγέλιο. Τώρα, ακούστηκε ένα σχόλιο για το μακροσκελή κατάλογο παρενεργειών των εμβολίων. Αντενδείξεων, συγγνώμη ε, όντως υπάρχει τέτοιος εκτενής κατάλογος και αυτό είναι το με τη συζήτηση που γίνεται για τον εμβολιασμό, οι αντενδείξεις. Μία αντένδειξη για κάποια εμβόλια είναι, και τον τρόπο παραγωγής τους, παρασκευής τους, είναι ότι όποιος έχει αλλεργία στα αυγά δεν θα πρέπει να κάνει το συγκεκριμένο εμβόλιο. Και ενδιαφέρουσες μελέτες απέδειξαν ότι πολλοί που έχουν αλλεργία στα αυγά δεν έχουν παρόλα αυτά αλλεργική αντίδραση και στο εμβόλιο. Βέβαια χρειάζεται η αρχή της προφύλαξης εδώ, να είμαστε επιφυλακτικοί και προσεκτικοί. Αυτά σημείωσα. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφος κατέγραψε περισσότερες ερωτήσεις και θέλει να συμπληρώσει. Ευχαριστώ καταρχάς για την πολύ ενδιαφέρουσα ερώτησή σας. Θα ήθελα να αρχίσω και από την ερώτηση της κυρίας Κάντενμπαχ, τι μπορούμε εμείς να κάνουμε στο Κοινοβούλιο, τι θέλετε από τους βουλευτές. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει το Κοινοβούλιο για την προώθηση των πολιτικών, για τον έλεγχο της εφαρμογής τους όχι μόνο στα κράτη-μέλη, βεβαίως είμαστε σε επαφή με τα κράτη-μέλη. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να υπάρχει δεδομένη η ε, πρόσβαση, ε, να είναι διαθέσιμα τα εμβόλια, να προβάλλεται αυτό, να φαίνεται και να βοηθήσουμε στην κατάσταση ε, την παρακολούθηση για να αντιμετωπίζουμε προβλήματα που μπορούν να αναδύονται συνεχώς για την κάλυψη και την αποτελεσματικότητα Δεν κάναμε διαφήμιση. Τι είπατε διαφημιστικό μήνυμα. Μια παρουσίαση κάναμε. Και ε, σας παρουσιάζουμε τα επιστημονικά δεδομένα. Uh, uh, ε, ε, όλα αυτά που λέμε τα βασίζουμε ε, σε ε, γερά επιστημονικά στοιχεία που κυκλοφορούν διάφορες φήμες για υποτιθέμενες παρενέργειες και τέτοια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να αναλύονται κάθε φορά. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει αποδειχθεί ότι αυτά είναι αβάσιμα. Απλούστατα θα πρέπει να τα κάνουμε στην άκρη και να σταματήσουμε να αναπαράγουμε κάτι το οποίο αποδεδειγμένα και πολλές φορές με μελέτες, αξιολογήσεις και εκτενώς έχει αποδειχθεί αβάσιμα διαβάσιμο ότι δεν συνδέεται ούτε με παρενέργειες ούτε με προβλήματα. Αυτό ισχύει για το ε, αλουμίνιο, ακόμα και για τον υδράργυρο. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Και εμείς στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχουμε κάνει μια αξιολόγηση για αυτά τα θέματα στο παρελθόν και καταλήξαμε με επιστήμονες, αξιόλογους, ανεξάρτητους που δεν έχουν καμία σχέση με φαρμακευτικές εταιρείε ή άλλα συμφέροντα. Αυτά δεν είναι καθόλου ε, στοιχειοθετημένα που κυκλοφορούν, είναι φήμες και καλό θα ήταν να σταματήσουμε να τα αναπαράγουμε. Και παρακαλώ όλοι να το λάβουμε υπόψη, διότι αν εμείς ζητούμε επιστημονικά στοιχεία και έρχεται η επιστήμη και σου λέει ότι αυτό δεν ισχύει, γιατί το συνεχίζεις, γιατί ζητάς επιπλέον επιστημονικά στοιχεία, τι άλλο να σου δώσει η επιστήμη από αυτό που σου έχει ήδη δώσει. Είναι φαύλος κύκλος από εκεί και πέρα και δεν πρόκειται να ξεφύγουμε ποτέ. Απλό είναι αυτό το ζήτημα. Άλλο θέμα για τις ανησυχίες σχετικά με την ε, Ουκρανία και τις ε, γειτονικές μας χώρες. Βεβαίως είναι σημαντικό το πρόβλημα και θα πρέπει να το παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά και η καλύτερη προστασία είναι να εξασφαλίσουμε εμβολιασμό ακριβώς για τις νόσους που προλαμβάνονται από τα εμβόλια. Για τις λοιπές δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να προστατεύουμε και τον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και να βοηθήσουμε και την ε, Ουκρανία και το λαό της Ουκρανίας να αυτοπροστατεύονται. Είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η κρίση. Και πάλι και για την Ελλάδα. Η ΠΟΗ έχει ένα πρόγραμμα συνεργασίας με την Ελλάδα τα τελευταία 4-5 χρόνια. Ε, τους βοηθούμε να αναθεωρηθεί το σύστημα υγείας, να υπάρξει κάλυψη όλου του πληθυσμού, πρόσβαση για τους πιο φτωχούς. Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, δεν είναι καθόλου εύκολα, αλλά Εξ όσων γνωρίζω από τα έργα αυτά και τα προγράμματα που έχουμε, έχει γίνει πρόοδος. Αξιόθαυμαστη τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως η κατάσταση γενικά ε, επηρεάζει και τα επιμέρους προβλήματα στην υγεία και δεν είμαι βέβαιος ότι τα αποτελέσματα αυτά θα είναι μόνιμα, αλλά έχουν γίνει προσπάθειες και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη και τη μετάδοση. Θα ήθελα απλώς ε, πρώτα απ' όλα να τονίσω και πάλι το εξής. Εμείς ξέρουμε ποια είναι η κάλυψη που ε, εξασφαλίζει την προστασία του πληθυσμού. Δεν είναι τυχαία αυτά τα στοιχεία. Ε, το 75% για το αντιγρυπικό θεωρείται στόχος. Αυτά δεν είναι ουρανοκατέβατα τα νούμερα, τα ξέρουμε, τα έχουμε ε, μελετήσει. Μπορούμε να κάνουμε και μια διάσκεψη για το 95% και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι στοιχειοθετημένα, υπάρχουν μελέτες. Δεν έχω ακούσει για παρενέργειες ή ανεπιθύμητες ε, όταν χρησιμοποιούνται πολλαπλά εμβόλια, ότι έχουν παρενέργειες ή ανεπιθύμητες ενέργειες. Ε, μπορεί κανείς να ανησυχεί για το κόστος, ας πούμε, αλλά η ανησυχία δεν έχει να κάνει με αυτό. Αλλά σκεφτείτε λίγο και το κόστος που θα προκαλούσε μια επιδημία ε, ε, εγκεφαλίτιδας από ε, αιμοφιλική γρήπη τύπου Β. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει και κόστος επιδημιών, δεν είναι μόνο του εμβολιασμού. Αυτά. Σταματώ εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ σύντομα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο συνάδελφος για το ρόλο των μελών του Κοινοβουλίου. Θεωρώ ότι ο εμβολιασμό ναι μεν είναι εθνική αρμοδιότητα και τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία καλούνται να εφαρμόσουν και να ε, αναπτύξουν και να οργανώσουν τον εμβολιασμό, αλλά ο ρόλος των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικός ε, στη χώρα του καθενό. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λαμβάνουμε αρκετέ γραπτέ ερωτήσει για του εμβολιασμού ζητούν κοινά προγράμματα εμβολιασμών ε, και ίσως και καλύτερο συντονισμό, αλλά δυστυχώς αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και τα, κράτη, και τα μέλη του Κοινοβουλίου έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Όσον αφορά το σχόλιο ότι δεν ε, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη στα σχόλια των πολιτών, ε, σαφώς και είναι πολύ σημαντικό ε, να λάβουμε σοβαρά υπόψη τους ε, πολίτες. Αλλά πρέπει να τονίσω ότι αυτό που χρειαζόμαστε εδώ είναι επιστημονικές ενδείξεις. Οι συνάδελφοι το, καλούν, ε, το αποκαλούν καλές, τεκμηριωμένες επιστημονικές ενδείξεις. Πρέπει να βασίζουμε τα πάντα σε συγκεκριμένες αποδείξεις. Αυτά έχω να πω ως προς αυτό. Όσον αφορά την Ελλάδα και εμείς έχουμε δραστηριότητες. Υπάρχει και η Επιτροπή ε, Ασφαλείας που ασχολείται με όποιο πρόβλημα προκύψει και προσφάτως υπήρξε και μια διαβούλευση με τα τέσσερα κράτη-μέλη που ε, πλήττονται περισσότερο από θέματα μετανάστευσης και ε, πρέπει να πω ότι τους βοηθήσουμε στην Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας να μπορέσουν ε, να ε, τα συνδυάσουν και με τα μέσα της πολιτικής ασύλου. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και σε αυτή την Επιτροπή, να δημιουργήσουμε κατάλληλους συνδέσμους με πολιτικές οι οποίες υπάρχουν σε άλλους τομείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι απαραίτητο στην υγεία, για παράδειγμα στη Γενική Διεύθυνση Home που υπάρχουν όλα αυτά τα κονδύλια για το άσυλο. Όσον αφορά τους λόγους για την έλλειψη εμβολίων, αυτή τη στιγμή είμαστε σε συζητήσεις με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τον EMA και οι συνάδελφοι στα αντίστοιχα τμήματα, στη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ, ε, προσπαθούν να έχουν μια συνολική εικόνα της κατάστασης και έχουμε πρόθεση να το συζητήσουμε και με τον κλάδο, να μας πούν για ποιο λόγο υπάρχει έλλειψη. Ε, είναι πρόβλημα παραγωγής, για παράδειγμα, ή πρόβλημα με τις προδιαγραφές που ισχύει σε κάθε κράτος μέλος. Ε, είναι κάτι το οποίο είναι εξελίξη αυτό. Ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό. Πριν ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση θα πρέπει να επανέλθω στο σημείο 17 γιατί ξέχασα να σας πω ότι οι συστάσεις των συντονιστών έχουν διανομηθεί δια της ηλεκτρονικής οδού και εάν δεν υπάρχει κάποια ένσταση θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας είναι στις 22 Ιουνίου. Έχουμε κοινή δημόσια κρόαση DEVE για τους στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους και η επόμενη συνεδρίασή μας στις Βρυξέλλες είναι στις 25 ε, Ιουνίου το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ. Πέρας της μακράς αυτής συνεδρίας. Σας ευχαριστώ.